Possiamo cominciare i nostri lavori. Vorrei prima di tutto darvi una buona notizia. Αρχίζουμε τη συνεδρίαση μας με μια καλή είδηση. Έχω μια νέα συνάδελφο, την κυρία Ντεγκρίπε, που αντικαθιστά το συνάδελφο Μπαρνιέ, που γίνεται επίτροπος. Εξ ονόματος όλων σας την καλωσορίζω και της εύχομαι καλή δουλειά στο Ευρωκοινοβούλιο και πιο συγκεκριμένα στην Επιτροπή μας. Ελπίζω να επιλέξει την Επιτροπή μας. Δυστυχώς έχουμε όμως και μία κακή είδηση. Χθες πέθανε η σύζυγος του συναδέλφου Μπουρλάνζ, που πολλοί από εσά ξέρετε. Ήταν ευρωβουλευτής από το 89 και πιο πριν ίσως, πάρα πολλά χρόνια. Σας το ανακοινώνω αυτό. Δυστυχώς ο θάνατος είναι η μοίρα όλων μας είναι ένα βαρύ πένθος. Παρότι θα μας πλήξει όλους κάποια στιγμή, θα μεταφέρω τα συλληπιτήρια όλων σας στο συνάδελφο Μπουρλάζ. Και ερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη. Καταρχήν πρέπει να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Αν δεν έχετε σχόλια ή παρατηρήσεις, θεωρούμε ότι εγκρίνεται. Ανακοινώσει του Πρόεδρου. Πρώτη, αποφασίστηκε να έχουμε μια άτυπη συνάντηση με εκπροσώπους της κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου του Βελγίου. Για να δούμε πώς θα γίνει αυτή η συνάντηση. Έχουμε επαφή με τις γερμανικές αρχές για να ξεκινήσει το πρόγραμμα που έχουμε αρχίσει να επεξεργαζόμαστε για πολιτικές και επιστημονικές συναντήσεις με εκπροσώπους των 27 χωρών μέσα στη διάρκεια της πενταετίας για θέματα που έχουν σχέση με την απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου που την έχουμε μελετήσει ήδη. Θέματα όπως το θέμα της εθνικής επικυριαρχίας της δημοκρατίας, της ταυτότητας. Πρέπει να μελετηθούν στα πλαίσια των σχέσεων μεταξύ κρατών και Ευρώπης. Ξέρετε ότι είχαμε πει οι πρώτες συναντήσεις να γίνουν στη Ρώμη και στο Βερολίνο. Η πρώτη συνάντηση καλό θα είναι να γίνει στο Βερολίνο γιατί ξεκινάμε από τις πολλές συζητήσεις και σχόλια που έχουν γίνει στο Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο. Μετά θα έχουμε και άλλες συναντήσεις. Πρώτα στην Ιταλία και μετά στην Ουγγαρία που θα πάρει τη σκητάλη ε, του Συμβουλίου από την Ισπανία. Επίσης θα ζητήσουμε μια συγκριτική μελέτη γιατί σε σχέση πάντα με αυτές τις συναντήσεις ως προς τις θέσεις των πρόσφατων αποφάσεων των συνταγματικών οργάνων η πάση των ανωτάτων δικαστικών αρχών της κάθε χώρας σε θέματα επικυριαρχίας, δημοκρατίας και ταυτότητας στα πλαίσια της ενσωμάτωσης στην Ένωση. Επίσης μια μελέτη για την ασφαλή χρήση τεχνολογιών με ηλεκτρονικές υπογραφές προκειμένου να ε, σε σχέση με θέματα όπου υπογράφουν ηλεκτρονικά πολίτες πρωτοβουλίες με βάση το άρθρο 11 της συνθήκης. Οι συγητές που ορίστηκαν με την σύμφωνη γνώμη των εισηγητών, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω τα ονόματα. Ο κύριος συνάδελφος Μέντες Δεβίγκο για τις δύο εκθέσεις σχετικά με τα προσωρινά μέτρα για τη σύνθεση του Κοινοβουλίου. Δηλαδή διαβούλευση για τη σύγκληση διακυβερνητικής διάσκεψης και συζήτηση για το αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση πρότασης να μη συγκληθεί συντακτική. Συνάδελφος Τσαρκόφσκι. Έκθεση για την αναγκαιότητα ή μη να προταθούν αλλαγές στον κανονισμό σχετικά με τις μονόπλευρες ενδεχόμενες δηλώσεις των κρατών μελών στα πλαίσια της έγκρισης μιας πράξης στο Συμβούλιο. Η ομάδα ΕΛΚ ζήτησε να οριστεί εισηγητής για τη διαδικασία του προπολογισμού 2011 και το μετασχηματισμό του συστήματο επιτροπολογία με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Αν ο συνάδελφο Μέντε Δεβίγκο θέλει να μα πει αν έγινε αυτή η επιλογή ή όχι. Μέντε Δεβίγκο στα αγγλικά. Ο κύριος Σαντάλγκας, κύριε Πρόεδρε, θα είναι εισηγητής του ΕΛΚ για το θέμα. Για την πρώτη έκθεση, εγώ είπα είναι δύο. Το ένα είναι η διαδικασία του προπολογισμού και η δεύτερη είναι μετασχηματισμό του της επιτροπολογία συνθήκη Λισαβόνα. Το ΕΛΚ νομίζω ζήτησε να οριστεί εισηγητής και για τις δύο αυτές, και για τα δύο αυτά θέματα Μέντες Δεβίγκο. Κύριε Πρόεδρε, σήμερα για τον προπολογισμό έχω το όνομα Σαλβάργας. Για το δεύτερο θα σκεφτούμε. Πρόεδρος. Ο συνάδελφος Σαοντάργας λοιπόν για τον προπολογισμό και για τη δεύτερη έκθεση θα περιμένουμε. Υπήρξε συμφωνία των συντονιστών στις 8 Φεβρουαρίου να οριστεί ο συνάδελφος Βέροφστατ εισηγητής για τη διαδικασία με συνδεδεμένες επιτροπές σχετικά με την σύσταση της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Το έχουμε συζητήσει ήδη. Είμαστε εισηγητές του πρώην άρθρου 50. Σημαντικός ο ρόλος μας. Η Επιτροπή Δημόσιων Ελευθεριών Μα ανακοίνωσε ότι σύντομα θα μελετήσει την πρόταση αλλαγή του κανονισμού σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα. Ελπίζω να συμφωνείτε ότι η πρόταση της Κομισιόν που υποβλήθηκε το 2008 με αρμόδια επιτροπή, την Επιτροπή Ελευθεριών, εισηγητής ο συνάδελφος Κάφμαν, η ΑΦΚΟ, για τα συνταγματικά δηλαδή, ε, παίρνει και αυτή με βάση το άρθρο 50 του κανονισμού με εισηγήτρια την κυρία Γετερμάκη. Ψηφίστηκαν οι τροπολογίες του Κάσμαν το Μάρτιο του 2009. Δεν ψηφίστηκε το νομοθετικό κείμενο ψήφισμα. Κατέπεσε το κείμενο και πρέπει να ξαναρχίσουμε από την αρχή τώρα πρέπει να ορίσουμε εισηγητή ή εισηγήτρια για γνωμοδότηση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Πάντως θεωρώ ότι συνάδελφος για τερμάκι δεν ξέρω πώς προφέρει για τερμάκι, για τερμέκι είπε ότι επιθυμεί να ε, αναλάβει και πάλι την αποστολή αυτή. Εγώ το θεωρώ λογικό το έτοιμο. Βέβαια, θα ακούσω τι έχουν να πούνε οι συναδελφοί. Έκθεση γνωμοδότησης. Βλέπω ο κύριος Ντάφ Καταφάσκη ε, και άλλοι εκπρόσωποι των ομάδων. Ωραία. Θεωρούμε ότι μπορεί η κυρία Αγιωταμάκη να είναι η Πρακτικά το συνεδριάσεων 18 Ιανουαρίου, 19 Ιανουαρίου, 25 Ιανουαρίου έχουν μοιραστεί. Αν δεν έχετε παρατηρήσεις, θεωρούνται ότι εγκρίθηκαν. κύριος Νταφ. Ε, νομίζω ότι δεν έχουν διανεμηθεί μέχρι στιγμής και χρειαζόμαστε ένα έγγραφο σχετικά με την ημερήσια διάταξη, το οποίο δεν έχουμε λάβει ακόμη, φαντάζομαι ότι είναι καθοδόν. Ε, βιάστηκα, λέει ο πρόεδρος. Η γραμματεία μου λέει ότι τα φορτηγά που μεταφέρουν τα έγγραφα από το Λουξεμβούργο δεν έφτασαν. Δεν ήρθαν. Βιάστηκα λοιπόν ότι, και είπα ότι μοιράστηκαν. Θα μοιραστούν πολύ σύντομα. Σημείο 5. Αναθεώρηση των συνθηκών με τα βατικά μέτρα όσον αφορά τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πολύ σημαντικό θέμα και επίγον. Δύο εκθέσεις. Η μία για το να μην συγκληθεί σύμβαση για την αναθεώρηση των συνθηκών και η άλλη ποια είναι αυτά τα μεταβατικά μέτρα. Θα τα συζητήσουμε από κοινού. Ζητήθηκε η γνώμη του Κοινοβουλίου από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από, τον, από πέρυσι ήδη με βάση το άρθρο του παράρτημα στη συνθήκη της Λισαβόνας και πρέπει να γνωμοδοτήσουμε και για την πρόταση του Συμβουλίου να μην συγκληθεί διακυβερνητική για τις ε, τροποποίησεις αυτές. Η συγητής Μέντες Δεβίγκο θα του δώσω αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως επενθυμίσατε, έχουμε δύο εκθέσεις δύο ψηφίσματα το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο τη Ολομελίας σε σχέση με το αίτημα το οποίο μας θέλει ο κύριος Βαν Ρόμπου, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σε επιστολή που απέστειλε στις 18 ε, Δεκεμβρίου στον πρόεδρό μας. Τι ερωτήσει είχε η επιστολή αυτή. Θα πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 48.3 της Συνθήκης, να συμφωνήσει αν θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συγκαλέσει μια διακυβερνητική και σε σχέση πάντα με το ίδιο άρθρο, εάν για αυτή την πρόταση αναθεώρησης της ε, συνθήκης στην οποία εγώ θα αναφερθώ, δεν χρειάζεται να συγκαλέσουμε και μία ε, convention, μία συνέλευση, όπως και στο παρελθόν. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσουμε αν όντω θα πρέπει να συγκληθεί και αυτή η συνέλευση εκτός από τη διακυβερνητική για την αναθεώρηση των συνθήκων. Πριν λοιπόν να δώσουμε σε αυτό το δεύτερο έτοιμο απάντηση, θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς περιέχεται στο σχέδιο ψηφίσματος το οποίο υπάρχει και γιατί μας ζητάει το Συμβούλιο τη δική μας εξουσιοδότηση για να συγκαλέσει ε, συνελεύσει συνελεύσεις αυτές τις δύο διαφορετικές, διακυβερνητική και την άλλη συνέλευση, την Convention. Όπως ξέρουμε, Ενάμιση μήνα σχεδόν μετά από τη θέση σε εσύ της Ειδικής Λισαβόνας, τι θέλει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να την τροπολπίσει. Ήδη, από τώρα. Για ποιο λόγο. Διότι η συνθήκη της Λισαβόνας ενεκρίθηκε, ακυρώθηκε με κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες, τις οποίες γνωρίζετε και δεν θα επαναλάβω, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό εμάς μας αφορά σε πρώτο λόγο, πρώτα απ' όλα, διότι μας αφορά η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο ρυθμός των βουλευτών. Και για μας αυτό είναι πολύ σημαντικό άμεσα. Για ποιο λόγο. Διότι προβλέπεται συνθήκη της Λισαβόνας, σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, φάση μιας έκθεσης την οποία εμείς εξετάσαμε, έκθεση των κυρίων Λαμασούρ και Σεβερίν που ε, τροπολογήθηκε εκ των υστέρων από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, προστέθηκε μία νέα έδρα, όπως ξέρετε, η οποία δόθηκε σε μία χώρα την οποία γνωρίζετε, αλλά η, συνθήκη της Λισαβόνας, βάσει της αρχή της αναλογικότητας, προβλέπει ένα άλλο σύστημα για την ε, αριθμό των εδρών κάθε χώρας. Θα πρέπει, λοιπόν, εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχουμε 751 συναδέλφους. Τι συνέβη. Δεν μπόρεσε η συνθήκη της Λισαβόνας, όπως ξέρετε, να τεθεί σε ισχύ έγκαιρα και να γίνουν οι τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές σύμφωνα με τις συνθήκες της Λισαβόνας. Έγιναν βάση της ε, συνθήκης της νίκης, που ήταν τότε η συνθήκη ισχύ. Έτσι λοιπόν έχουμε λιγότερους ευρωβουλευτές από αυτούς τους οποίους προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας. 736-751. Έχουμε λοιπόν μια διαφορά στον αριθμό των βουλευτών μεταξύ των δύο συνθήκων. Νίκαιας και ε, Λισαβόνας. Αυτό το είχε προβλέψει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο γνώριζε ότι δεν θα μπορέσει έγκαιρα να τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας. Η κατανομή που είχε γίνει Λοιπόν, τότε, ισχύει τώρα και δεν μπόρεσε να γίνει ακόμη η νέα κατανομή βάσει της συνθήκης Λισαβόνας. Έγιναν τα πράγματα με τις, παλ... συνθήκες που ίσχυαν στο παρελθόν. Και όπως ξέρετε υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των δύο συνδικών, διότι η Γερμανία χάνει τρεις βουλευτές και οι βουλευτές οι οποίοι εξελέγησαν με την συνθήκη της νίκαιας, δεν μπορεί τρεις μήνες μετά που τίθεται σε ισχύ μια άλλη συνθήκη να χάσουν τη θέση τους, να χάσουν την έδρα τους. Γι' αυτό θα πρέπει εμείς να πάρουμε μια απόφαση σχετικά με το θέμα αυτό. Και βεβαίως οι τρεις αυτοί συνάδελφοι, οι Γερμανοί που εξελέγησαν τον Ιούνιο, θα συνεχίσουν να είναι ευρωβουλευτέ μέχρι να τελειώσει η παρούσα θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτό μα ζητά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Να τροποποιήσουμε το πρωτόκολλο 36 υπόπτε τη ε, συνθήκη Λισαβόνα, ώστε να μπορέσει κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περίοδου να ε, διευθετηθεί το θέμα αυτό και συγχρόνως οι 18 βουλευτές οι περισσότεροι που προβλέπονται και δεν εξελέγησαν τον Ιούνιο να αποτελέσουν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τι μας λέει λοιπόν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα αλλάξουμε το πρωτόκολλο 36, θα προβλέψουμε ένα μεταβατικό καθεστώς ώστε να μπορέσουμε να προβλέψουμε τι θα γίνει με αυτούς τους καινούργιους 18 βουλευτές. Οι τρεις παραπάνω Γερμανοί θα ε, παραμείνουν ως το τέλος της θύρας τους και αυτό θα ισχύσει μέχρι να ολοκληρωθεί και η επόμενη ε, διακυβερνητική και να κυρωθούν και όλες αυτές οι αποφάσεις από τα 7 Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτό λοιπόν είναι μία μικρή ιστορική αναδρομή την οποία έκανα για να καταλάβετε περί ποιον στόχεται. Αυτό λοιπόν μα ζητά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και σύμφωνα με το σχετικό άρθρο τη συνθήκη, θα πρέπει εμεί να αποφανθούμε τώρα. Συμφωνούμε ή όχι με το αίτημα το οποίο μα έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στην πρόταση που σας υποβάλλω ή για να απαντήσω στο ερώτημα το οποίο ε, έστειλε το Συμβούλιο, δίδω καταφατική απάντηση. Σας προτείνω και προτείνω να προτείνουμε στην Ολομέλεια να εξουσιοδοτήσουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συγκαλέσει την διακυβερνητική διάσκεψη. Αυτό είναι το πρώτο θέμα του πρώτας ψηφίσματος που έχει μπροστά σας. Το δεύτερο θα ήθελα να πω. Θέλω να κάνω μια κριτική στο Συμβούλιο. Είμαστε σε μια κατάσταση κάπως ανώμαλη θα έλεγε, που δυσχεραίνει κάπω τα πράγματα και θα πρέπει να ανοίξει μια νέα διαδικασία κύρωση από τις 27 χώρε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να είχε διευθετηθεί διαφορετικά εάν το Συμβούλιο είχε πάρει σε εύθετο χρόνο τι αποφάσει που έπρεπε να πάρει. Δεν θέλω βεβαίω να αποκρύψω ότι με απασχολεί το εξής. Υπάρχει ένα κράτος μέλος, η Γαλλία, στην οποία η σύγκληση των εκλογών, των ευρωεκλογών, του πρασμένου Ιουνίου, δεν προέβλεπε την εκλογή των δύο συμπληρωματικών μελών που, προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας να δοθούν στη Γαλλία. Σε 11 χώρες λοιπόν, στην παρούσα κατάσταση δεν έχουμε δυσκολίες, αλλά στη Γαλλία υπάρχει πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, αυτό το λέει το Συμβούλιο και το λένε και οι γαλλικές αρχές, δεν υπάρχει τρόπος να εκλεγούν αυτοί οι δύο συμπληρωματικοί βουλευτές από τη Γαλλία. Ο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, προβλέποντας αυτή τη δυσκολία, σε προηγούμενες αποφάσεις, προέβλεψε το εξής. Και για αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, η γαλλική η Εθνική Συνέλευση της Γαλλίας να ορίσει, να ορίσει με εθνικές εκλογές, σε εθνικό μάλλον επίπεδο, συγγνώμη, πώς αυτοί οι δύο βουλευτές θα έρθουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάλιστα περιπτώσει, αυτό το άκουσα, είναι λεπτό το θέμα, θα το αποφασίσουν οι Γάλλοι. Απλώς θέλω να πω, όπως λέγω και στο σημείο 2 του σχεδίου απόφασης, ότι λυπούμε που έγιναν τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Κύριε Πρόεδρε, εμεί ακούσαμε την άποψη και του Συμβουλίου και ακούσαμε πριν από δύο εβδομάδες και την προηγούμενη εβδομάδα την Ισπανική Προεδρία να μας λέει ότι από νομικής πλευράς δεν υπάρχει άλλη λύση για να επιληθεί το θέμα εκτός αν γίνουν ε, στη Γαλλία νέες ευρωπαϊκές εκλογές για να εκλεγούν αυτοί οι δύο συμπληρωματικοί βουλευτές. Πράγμα το οποίο νομίζω ότι είναι απίθανο. Επίσης θα ήθελα να επενδύσω ένα άλλο θέμα κύριε Πρόεδρε. Ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την έκθεση Μάρτιν τον προηγούμενο Νοέμβριο που προεβλέπει οι βουλευτές αυτοί μέχρι να γίνουν πλήρη μέλη. Δηλαδή μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία βουλευτικής επικύρωσης να έχουν τη θέση και το καθεστώς του παρατηρητού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συμπεριλαμβάνονται εδώ και δύο τελειωτικές σκέψεις πάρα πολύ συμπληρωματικέ στην εκθεσή μου. Πρώτα απ' όλα, η οριστική απόφαση για την τελική σύνδεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να υποβληθεί και πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι τουλάχιστον προβλέπεται στους επόμενους, τα επόμενα χρόνια μία περαιτέρω διεύρυνση και ο κύριος Νταφ είναι εισηγητής της μιας έκθεσης για το θέμα αυτό στην Επιτροπή μας, άρα θα πρέπει να τονίσουμε εμείς ότι και στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε μία προσωρινή λύση για την τωρινή θητεία έως το 2014. Αλλά όταν θα ε, ληφθεί η οριστική απόφαση, θα πρέπει να μπορέσουμε να εγγυηθούμε ότι ο, αριθμός, ο τελικός αριθμός και ο οριστικός αριθμός των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι 751 βουλευτές. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω συμπερασματικά ότι νομίζω ότι πρέπει, εγώ προτείνω να εξισοδοτήσουμε το Συμβούλιο να συγκαλέσει την διακυβερνητική, λαμβάνοντας υπόψη ε, τις παρατηρήσεις που έκανε και πρέπει να πω ότι εμείς γνωμοδοτούμε θετικά. Δηλαδή, την εξουσιοδοτούμε το Συμβούλιο να την ε, συγκαλέσει αυτή την διακυβερνητική. Σχεδόν έχουν αποφασιστεί αυτά τα πράγματα, αλλά δεν ξέρουμε μέχρι τότε, μέχρι την τελική της σύγκληση, τι άλλα θέματα θα έχουν προκύψει. Αυτό το οποίο λοιπόν πρέπει να κάνουμε εμείς επαναλαμβάνω τώρα είναι να δώσουμε την εξουσιοδότησή μας για να μπορέσει να προχωρήσει η όλη η διαδικασία. Επίσης, άλλη επίπτωση του 48.3 και των νέων εξών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι το δεύτερο θέμα που περιλαμβάνεται στην έκθεση του κυρίου Βαν Ρόμπη. Για αυτή τη συγκεκριμένη αλλαγή χρειάζεται να συγκληθεί μία convention, μία νέα συνέλευση. Εγώ στην έκθεσή μου ανέλησα κάπως συνοπτικά το όλο θέμα, το οποίο γνωρίζετε ε, εσείς εξάλλου αρκετά καλά και πιστεύω ότι την, ε, τον τίτλο του σε άλλες αυτής της διάσκεψης, την Convention, εμείς εδώ την ε, εφήβραμε στο Κοινοβούλιο. Στην αρχή μιλούσαν για body, για κάποιο όργανο. Εν πάση περιπτώσει, εμείς για να μπορέσουμε να κάνουμε το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη και να κάνουμε την εκβαθέων μεταρρύθμιση ε, της, ε, του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, αν θέλετε, είπαμε ότι θα πρέπει να λέγεται αυτό το body convention. Εν λοιπόν, εφεύραμε τη λέξη αυτή, τη χρησιμοποίησαμε εμείς για πρώτη φορά και ξέραμε ότι ο στόχο τη είναι να μπορέσει να επιλύσει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που δεν έχει επιλυθεί. Και δεύτερον, ο χαρακτήρα τη είναι προσωρινό. Δηλαδή, κάποια μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην υπόλοιπη θητεία του Κοινοβουλίου. Μου φαίνεται όμως ότι δεν χρειάζεται να συγκληθεί και η Convention. Νομίζω ότι πρέπει να συγκαλείται τέτοιου είδους συνέλευση για σημαντικές μεταρρυθμίσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι πραγματικά ε, θέματα πολιτικής ε, σημασίας πλην των άλλων. Σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα δεν νομίζω ότι είναι μίζωνο σημασία το θέμα αυτό της σύγκλησης. Αυτή είναι λοιπόν η απόψή μου και ελπίζω θα είναι και δική της. Δεν είναι απαραίτητο να συγκληθεί και νέα convention και νέα συνέλευση για να επιληθεί αυτό το πρόβλημα σε αυτή την μεταβατική περίοδο και τη διάρκεια της υπόλοιπης παρούσας θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό είναι το περιεχόμενο των προτάσεων που εξ ονόματος της Επιτροπής υποβάλλω σε όλους εσάς και βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση ή σχόλιο. Είμαι ούτως ή άλλως στη διάθεσή σας και βεβαίως θα ακολουθήσω την άποψη της πλειοψηφίας όπως πάντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσασταν πολύ σαφείς. Όσον αφορά την πρόταση απόφασης για να δεχτούμε τη μη σύγκληση συντακτικής, θεωρώ ότι τα πράγματα είναι απλά. Πιο πολύ αξίζει να συζητήσουμε το δεύτερο θέμα τα προβλήματα της εισαγωγής των 18 νέων βουλευτών με σεβασμό τη συνθήκη που λέει όποιος εκλέγεται, εκλέγεται για πέντε χρόνια. Δεν μπορούμε να διώξουμε τρει Γερμανού από το Κοινοβούλιο. Πάσπως και για τα δύο θέματα αρχίζει η συζήτηση. Ποιος θέλει το λόγο. Νταφ πρώτος. Κύριε Πρόεδρε, Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Μέντες Λεβίγκο για την παρουσίαση που μας έκανε και νομίζω ότι πολύ σωστό έχουμε έναν Ισπανό εισηγητή στο θέμα αυτό διότι ε, Ξέρετε ότι υπάρχουν ε, τέσσερις βουλευτές από την Ισαπανία που θα προσθεθούν αν συμφωνήσουμε σχετικά με αυτή τη διαδικασία. Οπότε πολύ σωστό ε, είναι να έχουμε έναν ε, εισηγητή ο οποίος θα μας θα μας καλέσει στην τάξη εάν ξεφύγουμε από το στόχο μας. Άλλωστε η χώρα αυτή έχει τώρα την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και νομίζω ότι καλά θα ήταν να ρωτήσουμε ε, το Συμβούλιο εάν θα ήθελε επί του θέματος αυτού να κάνει να κάνει μία δήλωση ε, εξ ονόματος του κυρίου Βαν Ρομπόη, διότι εξετάζουμε τα θέματα αυτά της διακυβερνητικής με ε, την, μόνιμη, ε, τη μόνιμη προεδρία πλέον και όχι ε, την τριμερή προεδρία όπως στο παρελθόν. Επιπλέον, οι φιλελεύθεροι είναι πολύ ικανοποιημένοι με τις εξελίξεις και ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθούν γρήγορα καλό θα ήταν να ε, συμπέσουν με ε, την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών σε κάθε χώρα για την εκλογή των επιπλέον ε, ευρωβουλευτών κατά τρόπον ώστε να μην υπάρχουν διαφορές αναλόγως εθνικότητος αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να ε, είναι σε εφαρμογή των συνθήκων, διότι ξέρουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τις συνθήκες ή μάλλον να το αναδιαμορφώσω. Είναι δυνατόν να αλλάξουμε τις συνθήκες, αλλά ξέρουμε ότι αυτό ε, ορισμένες φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η Γαλλία μέχρι κάποιου σημείου θα έχει δύο εθνικούς βουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό είναι ένα τεχνικό θέμα. Εγώ όμως δεν το ερμηνεύω έτσι και μάλιστα εκπλήσωμαι. Πώς η Γαλλία δεν έχει προετοιμαστεί σωστά για να εκτελέσει μία απόφαση η οποία ελήφθη υπό την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από τον κύριο Σαρκοζή και από τη Γαλλία. Πώς είναι δυνατόν να επανερχόμαστε σε μία διαδικασία την οποία έχουμε ε, θεωρήσει ιστορικά σαν ε, ε, παρόμοια με τις μεθόδους του Ναπολέοντα Βοναπάρτη και αυτό την εποχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το να καθοριστούν λοιπόν δύο βουλευτές από άλλο κοινοβούλιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα θέσει προβλήματα σοβαρής συνταγματικής μορφής που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την δημοκρατική νομιμότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτό το λέω ότι δεν ενδιαφέρει πολύ μόνο εμάς, αλλά και τα εθνικά κοινοβούλια τα οποία στο τέλος θα πρέπει να ε, προσυπογράψουν αυτές τις αλλαγές των συνθήκων. Καλό λοιπόν θα ήταν να διαβουλευθούμε με τα εθνικά κοινοβούλια στα πλαίσια μιας ευρωπαϊκής συνέλευσης όπως αυτό έχει γίνει στο παρελθόν. Δηλαδή να συζητήσουμε από κοινού τα σοβαρά αυτά προβλήματα τα οποία προκύπτουν. Εγώ θα ήθελα η ε, ευρωπαϊκή αυτή συνέλευση να είναι περιορισμένου χρόνου και ε, συγκεκριμένου στόχου αλλά ε, να περιλαμβάνει τα σημεία τα οποία συνεφωνήθησαν το Δεκέμβριο στο σχέδιο των πρακτικών που προβλέπει την ε, παροδική ε, τοποθέτηση εθνικών βουλευτών ε, εις αυτό το Ευρωκοινοβούλιο οπότε η Γαλλία και οι άλλες εμπλεκόμενες χώρες θα έχουν δύο στόχους καταρχήν να να ξαναυπολογίσουν τα αποτελέσματα των περισσινών εκλογών ή ή να προβούν σε μερικές εκλογές, σε election παρσιέλ, για να μπορέσουν να καλύψουν αυτούς τους δύο βουλευτές από τη Γαλλία. Φοβάμαι, μάλλον με συγχωρείτε, είμαι υπερήφανος να πω ότι συμφωνώ στο πρώτο σημείο με τον ε, κύριο Μέντες Ντεβίγο αλλά εμείς ε, είμεθα υπέρ μιας ευρωπαϊκής συνέλευσης η οποία θα προηγηθεί ε, και, και μιας προκαταρκτικής διαβουλεύσεως προτού συγκληθεί αυτή η συνέλευση. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο τώρα ε, στην κυρία Γιαννάκου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, πράγματι το θέμα αυτό μοιάζει χωρίς προβλήματα, αλλά στην ουσία μπορεί να δημιουργήσει. Ήδη αναφέρθηκαν από τον κύριο Μέντες Δεβίγο ε, στην εισήγησή του, ε, γιατί το θέμα που τίθεται βέβαια είναι και η μεταβατική διάταξη που αφορά και στην υπέρβαση από τη συνθήκη της Λισαβόνας, που αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Δηλαδή, αν θεωρείται αυτό ε, αυτονόητο ότι η Γερμανία θα κρατήσει βουλευτές παραπάνω. Αυτό έχω την εντύπωση ότι είναι ένα θέμα που θέτει διάφορα ερωτηματικά. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτοί που έχουν εκλεγεί βεβαίως για μία πενταετία υπάρχει πρόβλημα και υπάρχει πρόβλημα σε ατομικό επίπεδο αλλά δεν ξέρω αν ε, σχετικά με το σύνολο και την ε, ε, θέση που πρέπει να έχουμε εμείς αφού θέλουμε πλήρη εφαρμογή και απόλυτη της Λισαβόνας είναι λογικό να κρατηθούν οι Γερμανοί συνάδελφοι εφόσον θα προσθεθούν άλλοι με βάση τη Συμφωνία της Λισαβόνας. Αυτό είναι το μόνο ερωτηματικό εγώ που θέτω. Κατά τα άλλα συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Μέντες Δεβίγο. Δεν νομίζω ότι πρέπει να συγκληθεί μια συνέλευση. Η συνέλευση συνεκλήθη για τα πολύ σοβαρά θέματα που αφορούσαν στις θεμελιώδεις ελευθερίες, συνεκλήθη για τη συνταγματική συνθήκη και πέτυχε τους στόχους της και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Για το ζήτημα αυτό νομίζω ότι πρέπει να συγκληθεί μια διακυβερνητική διάσκεψη η οποία θα λάβει βεβαίως υπόψη την άποψη του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κυρία Γιαννάκο. Ο έχει το Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Γεια σας, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα, εξ ονόματος της ομάδας μας, να πω το εξής. Η έκθεση του κυρίου Νόμνες Δεβίγκο ανταποκρίνεται στις πολιτικές θέσεις τις οποίες έχουμε για το θέμα αυτό. Δηλαδή, Πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε εκτός από τα πιο συγκεκριμένα θέματα τα οποία συζητήθηκαν, αναφέρθηκαν και στα οποία και εγώ θα αναφερθώ αργότερα, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ποιος είναι ο πολιτικός στόχος της έκθεσης αυτής και του ερωτήματος που τέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ έχουμε μία πολιτική συμφωνία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολύ πολύπλοκο. Αποτέλεσμα ισορροπιών που επιτεύθηκαν εδώ και πάρα πολύ ε, χρόνια που οδήγησαν σε χώρες να κάνουν κάποια πράγματα σύμφωνα με τη συνθήκη της νίκαιας και έγινε σύμφωνα με αυτή την συμφωνία κατανομής κάποια πράγματα. Ή είχαμε πει ότι τότε εξάλλου όταν θα έχουμε σύνταγμα στην Ευρώπη θα γίνουν οι απαραίτητε για να υπάρχει ισορροπία. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Να υλοποιήσουμε μία πολιτική συμφωνία που επέτυχαν οι 27 χώρες και που είναι συμφωνία μεταξύ όλων των 27 για την παρουσία μας στο Ευρωπαϊκό Συμβολίο. Και τι λέει αυτή η συμφωνία, ότι στην παρούσα θητεία θα έχουμε 18 συναδέλφους περισσότερους. Αυτή είναι η συμφωνία. Εξηγήθηκε πάρα πολύ σωστά στην παρούσα νομοθεσία ότι θα έχουμε 754, τρεις περισσότερους δηλαδή, για να μην ζημιώσουμε τη Γερμανία, σωστό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι 18 βουλευτές που αντιστοιχούν σε 12 χώρες που έχουν δικαίωμα να εκπροσωπηθούν με μεγαλύτερο αριθμό συναδέλφων εδώ, θα το υλοποιήσουν και θα ασκήσουν αυτό το δικαίωμα που έχουν. Άρα ποιο είναι το πρόβλημα το οποίο έχουμε εδώ. Να διευκολύνουμε και να κάνουμε επίσημη αν θέλετε μια πολιτική συμφωνία την οποία έχουμε επιτύχει μεταξύ μας και να εξασφαλίσουμε το δικαίωμα το οποίο έχουν οι 12 χώρες που δεν εκπροσωπούνται σωστά επί του παρόντος να εκπροσωπηθούν. Έτσι όπως τους αντιστοιχεί σύμφωνα με τη μία συνθήκη. Πρόκειται για 12 χώρες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που έχουν δικαίωμα να έχουν ένα, δύο, τρει, τέσσερι συναδέλφου περισσότερου μέχρι να φτάσουν στον ρυθμό που αντιστοιχεί στην πολιτική συμφωνία. Πρώτο πρόβλημα. Πώ θα εξασφαλίσουμε η πολιτική αυτή συμφωνία και το δικαίωμα αυτό να εξασφαλιστούν και να υλοποιηθούν. Και πιστεύω ότι για αυτό το θέμα η πρόταση που περιλαμβάνεται στην έκθεση του κ. Μέντε Δεβίγκο είναι λογική. Διότι αυτό το οποίο λέει είναι, ακούστε, δεν χρειάζεται να συγκαλέσουμε μια νέα συνέλευση η οποία θα ξαναρχίσει μια νέα πολιτική συζήτηση για να υλοποιηθεί μια πολιτική συμφωνία στην οποία έχουμε καταλήξει όλοι και με την οποία όλοι έχουμε συμφωνήσει. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πολύ λογική η απάντηση που έδωσε το Κοινοβούλιο στο Συμβούλιο λέγοντας ότι δεν χρειάζεται να συγκαλέσετε και τη συνέλευση. Συγκαλέστε την διακυβερνητική, μεταρρυθμίστε την συνθήκη μέσω της επιβεβαίωσης της συμφωνίας που έχετε. Θα κρατήσει δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία 5 λεπτά. Σε 5 λεπτά έχει λυθεί το πρόβλημα. Τι λέει λοιπόν το Κοινοβούλιο στο Συμβούλιο. Ενεργήστε με αυτόν τον τρόπο δεδομένου ότι επί τη ουσίας υπάρχει συμφωνία. Επίσης πρέπει να πω ότι πιστεύω ότι καλό θα είναι σε ένα από τα σημεία που προτείνει η έκθεση να πούμε ότι όσο διαρκέσει αυτή η διαδικασία επικύρωσης, γιατί ξέρουμε ότι η επικύρωση μπορεί να διαρκέσει μια ζωή, διότι δεν έχω καμία εγγύηση ότι 27 χώρες σύμφωνα με τα δικά του συνταγματικά συστήματα θα κάνουν σύντομα την επικύρωση και αν κάποιος δεν θέλει θα τρενάρει και δεν θα το κάνει και με αυτόν τον τρόπο θα καταστρατηγήσουν το δικαίωμα των 12 ε, χωρών να υλοποιήσουν μια συμφωνία πολιτική που έχει επιτευχθεί εδώ και καιρό. Λοιπόν, όσο διαδικεί όλη αυτή η διαδικασία κύρωση, και επαναλαμβάνω, μπορεί αυτή η όλη διαδικασία να διαρκέσει ένα, δύο ή τρία χρόνια, λέγει η έκθεση αυτή, μάλλον προτείνει, ότι καλό θα είναι να έρθουν αυτοί οι 18 συνάδελφοι Ω παρατηρητέ, χωρί δικαίωμα ψήφου, βεβαίω, χωρί δικαίωμα ψήφου, σωστό, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι αρκετά λογικό να τους δώσουμε την δυνατότητα, όπως έλεγε στην μεταρρύθμιση που κάναμε του κανονισμού, μουτάτης, μουτάντη, όπως έγινε και σε άλλες περιπτώσεις, να τους εξασφαλίσουμε το δικαίωμα των 18 συναδέλφων που χτυπάνε την πόρτα μας να μπουν μέσα. Τη δική μου τη χτύπησαν την πόρτα. Και όχι μόνο οι Ισπανοί, πολύ άλλοι συνάδελφοι. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να του δώσουμε τη δυνατότητα, χωρί δικαίωμα ψήφου, να συμμετέχουν στι εργασίε του Κοινοβουλίου. Διότι να ψηφίσουν ω παρατηρητέ δεν μπορούν. Τελείωσε. Λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο σωστά το εξήγησε ο κ. Νταφ. Όσον αφορά την φύση, αν θέλετε, τα χαρακτηριστικά αυτών των νέων βουλευτών. Δηλαδή, πρέπει όλοι ίσως να προέρχονται από ένα κοινό σύστημα εκλογικό. Συμμερίζομαι αυτό που λέει και μου φαίνεται, όπως λέγεται και στην έκθεση, ότι είναι λογικό να πούμε ότι είναι λυπηρό που μπορεί να προστρέξει σε διαφορετικό τύπο εκλογές μια χώρα μέσω μια τριπλής, αν θέλετε, εναλλακτική λύσης που συμφωνήθηκε πέρσι τον Ιούνιο. Εγώ είμαι υπέρ ότι όντως η έκθεση αυτή θα πρέπει να αναφέρει το ότι οι συνάδελφοι αυτοί θα πρέπει να προέρχονται από τους, από τους καταλόγους της 7ης Ιουνίου. Και μπορεί ίσω να το κάνει αυτό η Γαλλία, εάν μέσω νόμου προβλέψει κάτι που δεν το προέβλεψε και δεν το αποφάσισε τον Ιούνιο. Δηλαδή, να γίνει η εκλογή των δύο βουλευτών αυτών από την εκλογική λίστα των ευρωβουλευτών του Ιουνίου. Αλλά εδώ θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Δεν μπορούμε να αφήσουμε στα χέρια τους την υλοποίηση μία συμφωνίας έτσι όπως την αναφέρουμε. Τι θέλω να πω, ας το πω διαφορετικά. Δεν μπορεί μία χώρα με αυτά που κάνει να υποβάλει τις άλλες 12. Δηλαδή δεν μπορούν 12 βουλευτές να παραβιάσουν το δικαίωμα των υπολείπων 16 από 18. Πιστεύω λοιπόν ότι θα είναι σωστό και σοφό να πούμε στο συμβόλιο, Συμβούλιο το εξή. Μη συγκαλέσετε συνέλευση, δεν είναι ανάγκη. Συγκαλέστε την διακυβερνητική, μεταρρυθμίστε τη συνθήκη, αλλάξτε τον αριθμό των βουλευτών, προσθέσετε αυτούς τους 18 βουλευτές από τα 12 χώρες, ζητήστε από τις 12 χώρες να επιλέξουν αυτούς τους 12 και όταν ε, εγκριθεί η αλλαγή της συνθήκης, θα δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά ας μην κάνουμε κάτι το οποίο δύο άτομα κατά κάποιο τρόπο θα παραβιάσουν τα γενικότερα δικαιώματα των υπολείπων 18. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε και κατά την άποψή μου είναι παρκής η έκθεση αυτή είναι σωστή και νομίζω ότι θα πρέπει να την ψηφίσουμε κατά πλειοψηφία και να εγκριθεί ταχύτητα για να, ταχύτατα για να μπορέσει να προχωρήσει η όλη διαδικασία. Ευχαριστώ. Ε, Όπω ο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως σωστά επιχειρηματολόγησε ο συγητή μας Μέντε Δεβίγκο και ο Σνάφος Χαρεγκούι πριν από μένα, ο δρόμος μπροστά μας είναι υποχρεωτική κίνηση. Οι τρει Γερμανοί βουλευτέ έχουν πλήρε δικαίωμα να μείνουν στα πέντε χρόνια. Οι 18 έχουν δικαίωμα, όσο πιο σύντομα γίνεται, να αναλάβουν και αυτοί το έργο του. Και θα πρέπει, όπως προβλέπηκαν για τους 18 βουλευτές στις προηγούμενες εκλογές, Όσες χώρες δεν το έκαναν, γιατί δεν το έκαναν όλε οι χώρες, αυτό που έπρεπε να κάνουν είναι χρέο τους. Αυτό όμω το χρέος, αυτή η υποχρέωση, η παράγυψη δεν πρέπει να βαρύνει στην υποχρέωση της συνθήκης της Λισαβόνας όσον αφορά τον αριθμό των εδρών. Πρέπει λοιπόν να κινηθούμε προς την κατεύθυνση που μας δείχνει το Συμβούλιο. Πρέπει ουσιαστικά να συμφωνήσουμε δηλαδή με τη διαδικασία αυτή. Βέβαια, ας διευκρινίσουμε ότι μπορούμε να προσθέσουμε τα εξής δύο τεινά. Το ένα για τη γνωμοδότηση για τη διακυβερνητική. Είναι πέραν πάσης αμφιβολίας όπως είπε ο συνάφος Μέντες Δεβίγκο. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα μια συντακτική συνέλευση για ένα τέτοιο θέμα. Άρα να μην υπάρχει διακυβερνητική. Όμως Έχουμε και την πρόταση για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 36. Γι' αυτό θεωρώ το θέμα, το πρόβλημα μάλλον που έθεσε ο συνάδελφος Νταφ είναι υπαρκτό. Πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αλλά όχι όπως είπε ο συνάδελφος Νταφ, ως λύση. Έρχομαι στο θέμα που επισήμανε αυτός που μίλησε πριν από μένα, ο Ισπανός συνάδελφος. Δηλαδή, δεν συμφωνώ ότι μόνο η μόνη λύση για τη Γαλλία είναι ή νέε εκλογέ ή να ψαρέψει ένα βουλευτή από την Εθνική Βουλή. Και αυτό είναι που δεν με πείθει στις προτάσεις τροπολογιών του Συμβουλίου, τη τρίτη λύση ορισμού των βουλευτών. Το να γίνει μια ε, μέτρηση εξπόστ εκ των υστέρων τεχνικά δεν γίνεται και λόγω του γαλλικού εκλογικού συστήματος που αντίθετα με τον ευρωπαϊκό νόμο προβλέπει ε, όχι μία εκλογική περιφέρεια αλλά επιμέρους εκλογικές περιφέρειες στη Γαλλία. Διαφορετικά θα ήταν εύκολο να επιλέξουμε την άλλη λύση αλλά διότι επιπλέον νομικά από τη στιγμή που δεν έγιναν εκλογές που να ληφθεί υπόψη η εκλογή δύο επιπλέον βουλευτών, δεν μπορεί αυτό να γίνει εκ των υστέρων. Αυτό θα προσβληθεί στα δικαστήρια. Βέβαια, αυτό δεν αποκλείει το ενδεχόμενο τους δύο βουλευτές να τους πάρουμε μεταξύ των μη εκλεγμένων. Νομικά δεν είναι ένας νέος ορισμός των γαλλικών εκλογικών περιφερειών των 8 εκ των υστέρων είναι μια πολιτική λύση, ορισμός πολιτικός βουλευτών που έχουν ψηφιστεί από τους ε, πολίτες αλλά δεν εξελέγησαν. Πέρα από το τεχνικό θέμα των δύο πρώτων που έχουν το δικαίωμα αυτό, ως έχει το γαλλικό σύστημα αυτό βέβαια δεν είναι δυνατό να γίνει. Τι θέλω να πω, εμείς ως Κοινοβούλιο, αν συμφωνούμε με την γραμμή του Συμβουλίου, μπορούμε να πούμε ότι για το συγκεκριμένο αυτό σημείο υποδεικνύουμε έντονα την άλλη λύση. Να μην εκλεγούν μέσω της Εθνικής Βουλής, αλλά από υποψήφιους μη εκλεγμένους στα ψηφοδέλτια των ευρωεκλογών στη Γαλλία. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Βέβαια παραμένει το πρόβλημα και εκφράζω και εγώ τη γνώμη μου τώρα. Πρέπει να πούμε ποιες εκλογικές περιφέρειες ποιες θα είναι οι εκλογικές περιφέρειες, ποιοι πρώτοι, ποιες ε, εκλογικές περιφέρειες θα επιλέξουμε. Ο όχι αυτό που προτείνει η Γαλλία, το θέμα είναι να επιλεγούν δύο βουλευτές. Από τους δύο πρώτους μη εκλεγμένους από τις οχτώ εκλογικές περιφέρειες. Στο μέλλον βέβαια θα πρέπει ε, οι υποψήφοι όλοι να περνάνε από, τους, από τις λίστες για τις ευρωεκλογέ με καθολική ψηφοφορία. Συνεχίζουμε, λέει ο Πρόεδρος, με τον κύριο Βέροφστατ. Κύριε Πρόεδρε, <clears throat> καταρχήν ευχαριστώ όπως και οι άλλοι παρεμβαίνονται στον κύριο Μέντες Δεβίγκο για την έκθεση αυτή και θέλω να σας πω ότι ε, κάπως εκπλήσωμαι από την έλλειψη φιλοδοξίας. Στις 5-6 προτάσεις ε, ψηφίσματος τις οποίες διατυπώνει και στην ε, ιδέα που διατυπώνει να μην συγκαλέσουμε μία Ευρωπαϊκή Συνέλευση. Γιατί το τι πρόβλημα αντιμετωπίζουμε ε, είναι ε, μία πολιτική συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών που δεν προσυπόγραψε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή πρόκειται, από, πρόκειται για ε, ένα ερώτημα άλλων θεσμικών οργάνων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο οποίο μέχρι στιγμής ποτέ δεν ενεπλάκημεν επισήμως και ε, ουσιαστικά και ε, πρόκειται ε, για μία πολιτική συμφωνία η οποία έχει καταγραφεί σε πρακτικά και τώρα πρέπει εμείς πρέπει να διατυπώσουμε τη γνώμη μας σχετικά με την σύγκληση μίας Ευρωπαϊκής Συνελεύσεως και πώς αξιολογούμε μία τέτοια πιθανότητα δεν καταλαβαίνω λοιπόν διότι πρόκειται για αντιφάσεις. Από τη μια πλευρά λέμε ότι υπάρχει συμφωνία και πρέπει να επιταχύνουμε και από την άλλη πλευρά ότι ποτέ δεν πρόκειται να κυρωθεί αυτή η συμφωνία. Γι' αυτό και υπάρχουν οι μεταβατικές ε, διατάξεις που είναι αντιφατικές. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να εξετάσουμε εδώ είναι το συμφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει μία ε, περίπου αμυγός πολιτική ε, ε, αίτηση από την πολιτική αρχή να προσθέσουμε ευρωβουλευτές, αλλά ποιο είναι το συμφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εάν χρειάζεται να προσθέσουμε 10 ευρωβουλευτές ε, υπάρχουν ε, σημαντικές απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη λειτουργία του θεσμικού αυτού οργάνου και σαν παράδειγμα θα αναφέρω τη συζήτηση την οποία έχουμε ήδη κάνει και θα κάνουμε στο μέλλον στις διασυνοριακές ε, λίστες όπου υπάρχει μία συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών που θα ήθελαν το 2014 να υπάρχουν πραγματικές ευρωπαϊκές εκλογές και όχι και καλυμμένες εθνικές εκλογές για να μπορέσουμε να αυξήσουμε την ε, ε, νομιμότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διότι ε, εάν ε, πρόκειται να συγκληθεί μία Ευρωπαϊκή Συνέλευση για να επικυρωθούν 18 ε, ευρωβουλευτές οι οποίοι δεν έχουν εκλεγεί αμέσως δεν μπορούμε εμείς να πούμε ότι αν γίνει όλη αυτή η φασαρία, όλη αυτή η δουλειά εάν γίνει μία Ευρωπαϊκή Συνέλευση γιατί δεν μπορούμε να προσθέσουμε άλλα αιτήματα, άλλες μεταρρυθμίσεις, άλλες προτάσεις για απαιτήσει που εμείς έχουμε έναντι των εθνικών ε, κοινοβουλίων ε, και μπορούμε να αναφέρουμε διάφορα παραδείγματα όπως παραδείγματο χάρη στις διασυνοριακές ε, λίστες για το 2014 σε επόμενες ευρωεκλογές. Οπότε τα θέματα αυτά θα αντιμετωπιστούν τελείως διαφορετικά. Δεν μιλάμε εδώ για μία μικρή συνέλευση δεν θα, σε ένα τέτοιο όργανο δεν θα ασχοληθούμε μόνο με τους 18 ευρωβουλευτές αλλά με όλα τα μεγάλα θέματα οπότε είναι το κατάλληλο σημείο να συγκληθεί μια τέτοια συνέλευση για να συζητηθούν αυτά τα σοβαρά θέματα. Διότι την πρώτη φορά όταν έγινε η πρώτη συνέλευση στο Λάκεν, στη διακήρυξη του Λάκεν, όπου ήταν μία πρόταση την οποία υπέβαλε ο πρόεδρος του Συμβουλίου εκείνη την εποχή και τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενθουσιάστηκε τώρα που προβλέπεται μία συνέλευση ε, σαν δυνατότητα στο, στη συνθήκη αντιδρούμε. Το όταν δεν υπήρχε και το πρότεινε το Συμβούλιο ενθουσιάστηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα που προβλέπεται ή στα θεσμικά όργανα ότι μπορεί να οργανωθεί κάτι τέτοιο τότε λέμε ότι δεν είναι αρκετά σοβαρό. Λοιπόν, πρότασή μου είναι να φροντίσουμε αυτή η διακυβερνητική συνέλευση να καταστεί σημαντική για να μπορέσει να γίνει μια Ευρωπαϊκή Συνέλευση και να ζητήσουμε από το Συμβούλιο να προσθεθούν και θέματα που ενδιαφέρουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως παραδείγματο χάρη οι διασυνοριακές λίστες πράγμα το οποίο θα αυξήσει το δημοκρατικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πιστεύω κύριε Πρόεδρε ότι την επόμενη φορά θα πρέπει να το συζητήσουμε και ε, να συζητήσουμε και για πιθανές ε, αλλαγές ε, εις ε, το, στις τροπολογίες και για να συζητήσουμε όλες τις τροπολογίες που θα τεθούν σχετικά με τις δύο εκθέσεις που ακούσαμε σήμερα. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Σταρκόφσκι. Καταρχήν, θα είμαι, ε, θα είμαι ειλικρινής, θα μιλήσω ανοιχτά και ίσως ε, και απλά. Υπάρχουν δύο θέματα, ένα θέμα αρχής και ένα θέμα ε, πιέσεως προς το Συμβούλιο σχετικά με τι εναλλακτική λύση θα προτιμήσουμε και ποιους βουλευτές θέλουμε να στείλουμε. Αλλά πολλοί είπαν ότι το να υπάρξει μία συνέλευση ευρωπαϊκή για να ασχοληθεί μόνο με αυτό το θέμα ε, ε, είναι υπερβολή αλλά απ' την άλλη προευλά μπορεί να δημιουργήσουμε ένα προηγούμενο που δεν θα μας αρέσει. Λοιπόν, όταν μιλάμε για νέους ευρωβουλευτές έχουμε και άλλο πρόβλημα ότι τι είναι πιο σημαντικό η νομιμοποίηση ή η εκπροσώπηση διότι όταν μιλάμε για νομιμοποίηση η γαλλική κυβέρνηση μας ζητά να δεχθούμε δύο βουλευτές από το Εθνικό Κοινοβούλιο τους από την άλλη πλευρά όμως θέλουμε αυτό το κοινοβούλιο να εκπροσωπεί όσο το δυνατόν περισσότερο τους πολίτες και όσο το δυνατόν δυνατόν πιο γρήγορα τους πολίτες. Υπάρχουν τα δύο αυτά θέματα. Εάν δεν γίνει λοιπόν μια τέτοια συνέλευση, το Συμβούλιο μπορεί να δεχθεί την άποψή μας, δηλαδή ότι δεν είναι δυνατό να δεχθούμε την τρίτη λύση. Και εδώ έρχομαι στο συμπέρασμα, δηλαδή με τι σειρά θα προχωρήσουμε. Εάν όλοι συμφωνήσουμε ότι δεν δεχόμαστε την τρίτη εναλλακτική λύση και αυτό θα πρέπει να είναι προσυμπεφωνημένο, τότε είναι σαν ε, να στέλνουμε το μπαλάκι στο Συμβούλιο και να περιμένουμε την αντίδρασή τους. Εάν ε, πούμε ότι δεν θα συγκαλέσουμε γρήγορα μία συνέλευση, δεν έχουμε καμία πίεση προς το Συμβούλιο. Εάν λοιπόν εμείς δεν αποφασίσουμε σε ε, δύο εβδομάδες ή σε ένα μήνα μπορούμε να στείλουμε το μπαλάκι στο Συμβούλιο και να τους πούμε ότι δεν δεχόμαστε την τρίτη εναλλακτική λύση. Όλοι όμως θα πρέπει να έχουμε συμφωνήσει ότι είναι απαράδεκτη η τρίτη εναλλακτική λύση και να έχουμε αποφασίσει τι μας ενδιαφέρει περισσότερο η νομιμοποίηση ή η εκπροσώπηση διότι αν θέλουμε να είναι αντιπροσωπευτικό το Ευρωκοινοβούλιο ως το δυνατόν πιο γρήγορα πρέπει να κατατάξουμε τα πράγματα με μια συγκεκριμένη σειρά πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε καταρχήν περί της πρωτής της σημασίας της εκπροσώπησης ή της νομιμοποίησης Συμφωνώ ότι εάν συγκληθεί ε, μία συνέλευση για αυτό το θέμα θα υποβαθμίσουμε τη σημασία του θέματος αυτός προς ε, όλη την εκλογική βάση πράγμα που δεν είναι προς συμφέρον μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φόξ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Τεβίγκο για την έκθεσή του και συμφωνώ με τα πορίσματα του. Δεν συμφωνώ με τον κύριο Βεροστάτη. Χαίρομαι για το ότι δεν υπάρχει μεγάλη φιλοδοξία. Γιατί όταν οι φιντεραλιστές που κάθονται μπροστά μου όταν αρχίσουν να μιλάνε για φιλοδοξίες εγώ τρομάζω. Γιατί αναπόφευκτα αυτό σημαίνει να αφαιρεθούν εξουσίες από τα εθνικά κράτη. Και όπως είπε επειδή ανάφερε στις υπερεθνικές λίστες ο κύριος ε, Βερόφστατ, εγώ το θεωρώ αυτό απέσιο. Θεωρώ ότι θα μειώσει τη δημοκρατική νομιμότητα και θα αυξήσει την προοπτική οι εξτρεμιστές να πάρουν περισσότερες έδρες στο Ευρωκοινοβούλιο. διοδός, οι τρεις Γερμανοί βουλευτές θα πρέπει να παραιτηθούν ταυτόχρονα με τους 18 επιπλέον βουλευτές που θα έρθουν εδώ. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι η απόφαση αυτή απαιτεί ομοφωνία. Άρα είναι πολύ πιθανό η γερμανική κυβέρνηση να μην συμφωνήσει με την πρόταση αυτή. Μέχρι το 2014 να φύγουν δηλαδή, να μην φύγουν, να ζητήσει να μην φύγουν οι τρεις Γερμανοί. Οπότε θα υπάρξει πρόβλημα με τους 18 υπόλοιπους. Αν οι Γερμανοί κρατήσουν τους επιπλέον βουλευτές τους τρεις μέχρι το 2014, το τίμημα είναι μικρό. Α του κρατήσουμε προκειμένου να έχουμε σύντομα του επιπλέον 18. Για να οριστούν αυτοί οι 18, το πώ θα γίνει αυτό, α το αφήσουμε στα κράτη-μέλη να το αποφασίσουν. Μην παρεμβαίνουμε εμείς. Είναι δικό τους δικαίωμα να επιλέξουν ποιο θα εκπροσωπεί το έθνο του. Ευχαριστώ. Πρόεδρο. Τιν ή τάιν η συνάδελφος. Τάιν λέγομαι κύριε Πρόεδρε. Το όνομά μου είναι Τάιν. Κάπως εξεπλάγει όταν διάβασα προηγουμένως την έκθεση ότι δεν είναι υποχρεωτική μία συνέλευση διότι αυτό είναι ένα θέμα που έχει συζητηθεί επανειλημμένως και εδώ είμαστε στο θέμα της ε, συγκροτήσεως ε, του Ευρωκοινοβουλίου αλλά είχαμε συζητήσει ε, το θέμα της συνέλευσης και είχαμε απορρίψει την ιδέα ότι μπορούν οι δύο Γάλλοι να καθοριστούν από το Εθνικό τους Κοινοβούλιο. Βέβαια η σύγκληση ε, μια συνελεύσεως κρατά πολύ καιρό και εντωμεταξύ δεν θα μπορέσουν ε, να προσέλθουν οι 18 ευρωβουλευτές. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει πλήρης ισοτιμία των εκλογών. Πρέπει οι εκλογές αυτές να είναι ίσες παντού ε, και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να εξισώσει το Ευρωκοινοβούλιο με τα εθνικά κοινοβούλια Τώρα αν πρόκειται για μία ή δύο ψήφους θα σας πω ότι όταν μιλούσαμε για την ελευθερία του τύπου στην Ιταλία η διαφορά ήταν μία ή δύο ψήφους. Άρα μπορεί να είναι κρίσιμες οι ψήφοι αυτοί, ε, ίσως όχι υποχρεωτικά προς την κατεύθυνση που θέλουμε. Είναι επίσης θέμα ενός προηγουμένου που θα δημιουργηθεί. Διότι αν δημιουργηθεί προηγούμενο τότε και στο μέλλον θα είναι δυνατόν να αποφασίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή ε, θα θυμάστε ότι είχαμε αλλάξει τις συνθήκες και στο παρελθόν. Είχαμε, μία, ε, ε, είχαμε εκλογές και μετά κυρώθηκε η συνθήκη. Δηλαδή το πρόβλημα θα προκύπτει και στο μέλλον. Πρέπει να σκεφτόμαστε μπροστά και να συμφωνήσει το Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και δεν θα πρέπει ε, γρήγορα ε, και στο πόδι να λάβουμε μία τέτοια απόφαση εκτός και αν μας πούν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Μέχρι στιγμής δεν κατάλαβα παρόλες τις δηλώσεις που έχουν γίνει γιατί η Γαλλία δεν μπορεί να προσθέσει αυτούς τους δύο εθνικούς βουλευτές. Δηλαδή το ακούω αλλά δεν ξέρω τι γίνεται η Γαλλία. Ήξερε πάρα πολύ καλά ότι θα έχει δύο επιπλέον ευρωβουλευτές όταν θα ισχύσει η συνθήκη της Λισαβόνας πρώτων των ελευταίων εκλογών. Οπότε είπε, έπρεπε να έχουν λάβει τα μέτρα τους επ' αυτού. Οπότε σε περίπτωση ανάγκης θα πρέπει ίσως η Γαλλία να μην έχει αυτούς τους δύο ευρωβουλευτές στη μεταβατική φάση μέχρι ότου μπορέσουν να συναποφασίσουν και οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ και το λόγο έχει τώρα η κυρία Ντερίντ η οποία ενδιαφέρεται γιατί είναι Γαλλίδα. Καταρχήν σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια που με καλωσορίσατε. Η πρώτη μου παρέμβαση στην Επιτροπή των Συνταγματικών Θεμάτων δηλώνω τη μεγάλη μου χαρά που είμαι Ευρωβουλευτής και που θα μπορώ να παίρνω μέρο στις εργασίες της Επιτροπής Συνταγματικών Θεμάτων. Θα περιοριστώ μόνο στο γαλλικό θέμα. Γιατί το το θέμα αυτό σχολιάστηκε αρκετά από αυτούς που μίλησαν πριν από μένα. Θα ήθελα να σα δώσω μερικά πληροφοριακά στοιχεία και διευκρινήσει. Όντω, στη Γαλλία οι Εθνικέ αρχέ έχουν επιλέξει την τρίτη λύση. Μία από τι τρει λύσει. Εκλογές ad hoc ήταν η μία να ληφθεί υπόψη τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών του Ιουνίου 2009 και τρίτον ορισμός από το Εθνικό Κοινοβούλιο <coughs> βουλευτών για να γίνουν ευρωβουλευτέ. Η τρίτη λύση επελέγει από την κυβέρνηση. Η λύση υπαριθμών 3 που σημαίνει η Γαλλία θα αφήσει η Βουλή όπου οι βουλευτές έχουν εκλεγεί με καθολική ψηφοφορία η Βουλή θα συνεδράσει σε Ολομέλεια και θα εκλέξει δύο βουλευτές να σταλούν στο Ευρωκοινοβούλιο. Στην αρχή ως παρατηρητές και όταν θα επικυρωθεί το πρωτόκολλο από όλες τις χώρες τα δύο συγκεκριμένα άτομα που θα έχουν επιλεγεί, εκλεγεί αν θέλετε από την Εθνική Βουλή αμέσως θα καταθέσουν την εθνική εντολή και θα γίνουν ευρωβουλευτές πλήρης. Τακτικά μέλη. επιφανής νομικοί, συνταγματολόγοι στη Γαλλία βοήθησαν την κυβέρνηση να επιλέξει την λύση 3. Γιατί έγινε αυτό, διότι αυτή η λύση είναι η μόνη οι οποίοι δεν συναντά νομικά και συνταγματικά εμπόδια, ανυπέρβλητα. Η πρώτη λύση, εκλογή ad hoc, που πρώτον θα ήταν εκλογή που θα στοιχήσει πάρα πολύ και θα είναι περίπλοκη και δεν θα ενδιαφέρει ιδιαίτερα, συγκινήσει ιδιαίτερα τους εκλογής Και υπάρχει ένα πρόβλημα επιπλέον. εκλογής περιφέρειας οι δύο βουλευτές που ενδεχομένως θα έβγαιναν από μια εκλογή αναπληρωματική ας την πούμε, ad hoc, θα εκπροσωπούσαν θα, θα είναι διαφορετικοί από τους 72 άλλους Γάλλους ευρωβουλευτές που προέρχονται από συγκεκριμένες εκλογικές περιφέρειες. Διότι αν έχουμε εκλογές αναπληρωματικές ad hoc, επί τούτου οι δύο βουλευτές δεν θα βγαίνουν από περιφερειακή εκλογική περιφέρεια, θα προέρχονται από μια ευρωπεριφέρεια της Γαλλίας. Και αυτό δημιουργεί de facto μια στρέβλωση, μια ανισομέρεια ανάμεσα στην εκλογική περιφέρεια από την οποία θα προέρχονται και τους 72 άλλους Γάλλους ευρωβουλευτές που έχουν εκλεγεί σε περιφερειακή βάση. Και δεν είναι δεν θα υπάρχει σημαντική ευρωπαϊκή διάσταση στην περίπτωση αυτή που θα κινητοποιούσε τους Γάλλους εκλογής αν κάναμε αναπληρωματικές εκλογές σε όλη τη Γαλλία για να εκλεγούν δύο επιπλέον Γάλλοι ευρωβουλευτές. Η δεύτερη λύση. Να αναχθούμε στις εκλογές του Ιουνίου του 2009. Τη μελέτησαν και αυτή τη λύση οι νομικοί στη Γαλλία εδώ υπάρχει πρόβλημα βάσης. Δηλαδή, πού στηρίχθηκε, τι είδους απογραφή αποτέλεσε τη βάση για τις δύο επιπλέον έδρες και πώς θεωρηθούν οι περιφερειακές εκλογικές περιφέρειες για τους δύο αυτούς επιπλέον ευρωβουλευτές. Όπως ξέρετε, μάλλον, οι ευρωεκλογέ του Ιουνίου 2009 έγιναν με βάση την απογραφή του 2006. Αυτά είναι τα τελευταία γνωστά νούμερα. Απογραφή πληθυσμού 2006. Και μοιράστηκαν τα νούμερα αυτά στις 8 περιφέρειες. Από τότε μέχρι σήμερα έγινε και άλλη απογραφή του 2007. Και έχουμε τα νούμερα της απογραφής του 2007 που είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα τη δημογραφική πραγματικότητα της Γαλλίας. Άρα και των εκλογέων σε σχέση με τον Ιούνιο του 2009. Ποια, θα, ποια απογραφή θα είναι η βάση. Για τη δεύτερη λύση. Θα στηριχτούμε στην απογραφή του 2006 αλλά υπάρχουν και πολλά επιχειρήματα που συνηγορούν, που δεν συνηγορούν υπέρ της λύσης αυτής. Γιατί, όπως σας είπα, στο μεταξύ έχουμε τα νούμερα της απογραφής του 2007. Για να είμαστε πιο κοντά στην πραγματικότητα του ολοκληρωτικού στόματος να στηριχτούμε στην απογραφή του 2007, που είναι διαφορετική από τη βάση για τις εκλογές του 2009 για το ποιες από τις 8 περιφέρειες θα πάρουν τους δύο ευρωβουλευτές και ανάλογα με το ποιο θα πάρουμε μας βάση, αν πάρουμε τα νούμερα από γραφή 2006 ή τα νούμερα από γραφή 2007, τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά. Και η μία και η άλλη λύση επιδέχονται αμφισβήτηση. και θα μπορούσαν να γίνουν προσφυγές, να αναζητηθούν επιχειρήματα υπέρ ή κατά και των δύο λύσεων. Στο όνομα υπόνοιας, υποψίας, ε, ότι η επιλογή εκ μέρους των γαλλικών αρχών για την α ή την β βάση ότι θα οδηγούσε στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Θα μπορούσε να υπάρξει σοβαρή αμφισβήτηση και αυτό θα αποδυνάμενε και το σύστημα και γενικά την ισχύ εκλογής αυτών των δύο βουλευτών. Τώρα ένα άλλο ερώτημα. Γιατί η Γαλλία δεν το πρόβλεψε αυτό. Τους δύο επιπλέον ευρωβουλευτές που θα τους έπαιρνε με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ειλικρινά δεν νομίζω ότι μπορούμε να το θεωρήσουμε αυτό αμέλεια ή παράληψη ή επιπολαιότητα οι πιο έγκριτοι συνταγματολόγοι Γάλλοι σοβαρά έκουρσαν τον κόδωνο του κινδύνου για την κυβέρνηση ως προς το εξής. Το Γαλλικό Σύνταγμα και η νομολογία και οι αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου από ό,τι φαίνεται δεν επιτρέπουν την εγγραφή σε εκλογικό νόμο άρθρου που να εξετάται από την ενδεχόμενη ισχύ μιας συνθήκης που δεν έχει ακόμα επικυρωθεί από όλου τους συνυπογράφοντες. Υπάρχει δηλαδή μια δυνητική ρήτρα που θα απαγόρευε κάτι τέτοιο. Και αυτό αποδυναμώνει έναν εκλογικό νόμο που θα στηριζόταν σε ένα τέτοιο δυνητικό όρο. Και οι νομικοί και οι συνταγματολόγοι στη Γαλλία που συμβούλευσαν τη γαλλική κυβέρνηση επέστησαν την προσοχή της κυβέρνησης στον κίνδυνο αντισυνταγματικότητας μιας τέτοιας κίνησης. Με αυτά τα δεδομένα επεδείχθη πνεύμα ρεαλισμού. επιλέγει η λιγότερο κακή λύση. Εκλογή από τη Γαλλική Βουλή, η οποία Γαλλική Βουλή μην ξεχνάμε, εκλέγονται τα μέλη με καθολική ψηφοφορία. Η λύση αυτή φαίνεται να είναι η καταλληλότερη προκειμένου να αποφύγουμε κινδύνους αμφισβήτησης του αποτελέσματος και της απόφασης συνταγματικού χαρακτήρα. Εξάλλου τα μέτρα αυτά είναι μεταβατικά και οι Γάλλοι βουλευτές που θα εκλεγούν, που θα έχουν ήδη εκλεγεί στη, έχουν εκλεγεί στην Γαλλική Βουλή, από που θα επικυρωθεί το πρωτόκολλο, θα καταθέσουν την εθνική εντολή για να γίνουν ευρωβουλευτές. Υπήρξε βούληση ρεαλισμού, χάραξης του λιγότερο επικίνδυνου δρόμου έτσι ώστε να αποφύγουμε ενδεχόμενε ενστάσεις, πράγμα που θα μπλοκάριζε τα πράγματα για πάρα πολύ καιρό, ρεαλισμός. Επελέγει η λιγότερο κακή λύση. Θεώρησα σκόπιμο να κάνω αυτές τις παρατηρήσεις αφού άκουσα τα σχόλια των συναδέλφων και θα εξακολουθήσω να παρακολουθώ τη συζήτηση με μεγάλο ενδιαφέρον. Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε. Ο συνάδελφος Σούλτς ζήτησε το λόγο. Σόλτς. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είναι ένα ουσιαστικό πρόβλημα με το, το οποίο αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή και επειδή είμαι νεοφερμένος στην Επιτροπή αυτή δεν θέλω να επισέλθω σε πολλές λεπτομέρειες συμφωνώ όμως με τον συνάδελφο Φερχόφστατ όταν λέει ότι πρέπει να εξετάσουμε ουσιαστικά το θέμα των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Νταφ να ε, επιταχύνει τις εργασίες του στο σχετικό θέμα διότι χρειαζόμαστε ε, λίγο χρόνο. Δεν όμως κάτι καινούριο. Θυμάμαι το, ε, τι συνέβη με τους ε, ε, ανατολικογερμανούς ευρωβουλευτές οι οποίοι στην αρχή ήταν παρατηρητές μέχρι σότου ε, ε, να μπορέσουν να εκλεγούν μετά από τις ε, εθνικές εκλογές που έγιναν μετά την επανένωση των Γερμανιών και επέτρεψε να έρθουν και οι σχετικοί ευρωβουλευτές από τη Γερμανία εδώ. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε το σχετικό άρθρο και να πούμε ότι ε, για αυτή ε, την μεταβατική περίοδο όταν δεν είναι έτοιμη μία χώρα και δεν έχει επαρκής ε, ευρωβουλευτές να μπορέσει να διαθέσει δύο εθνικούς βουλευτές. Δεν πρόκειται μόνο για νομιμότητα αλλά και για συμβολισμό διότι με την, ε, ε, την ισχύ της ε, συνθήκης της Λισαβόνας αναβαθμίζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο την, προσκήνιο για να προασπιστεί τα ενδιαφέροντα των πολιτών και ασχέτως πόσο φτάσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούμε πλέον να εμπλακούμε στην Ευρωπαϊκή Πολιτική πολιτική. Οπότε στα πλαίσια αυτά νομίζω ότι η ιδέα της συνέλευσης είναι ίσως υπερβολική για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά ε, εάν πρόκειται απλώς ε, ε, για ε, την, τον καθορισμό ευρωβουλευτών αλλά θα πρέπει να ξαναεξετάσουμε το θέμα γιατί αυτά τα οποία συζητάμε εδώ είναι πολύ σημαντικά για μία αύξηση της συμμετοχής και της επιρροής των πολιτών στα 27 κράτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και στην επόμενη, σε επόμενες θα πρέπει να συζητήσουμε και το θέμα αυτό διότι πολλές φορές μας λένε μετά τις εκλογές ότι οι ε, ε, πολίτες δεν εμπιστεύονται πλέον τους ευρωπαϊκούς θεσμούς αλλά εμείς πρέπει να τους ε, δώσουμε και πάλι εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό σύστημα. Ευχαριστώ. η κυρία Γκουρμάη. Ας δούμε καταρχήν τα γεγονότα. Καταρχήν Ε, είχαμε στην αρχή μη 751 ευρωβουλευτές και μία μεταβατική περίοδο. Το ερώτημα είναι ε, τι χρόνο θα καλύψει η μεταβατική περίοδο. Γνωρίζουμε ε, τους ευρωβουλευτές, θα θέλαμε να προσέλθουν να μπορέσουμε να αρχίσουμε τη δουλειά μας και όλα αυτά προβλέπονται στην κύρωση των ε, ε, εγγράφων ε, γιατί προσωρινά μπορούν μόνο να είναι παρατηρητές. Δεν υπάρχει μία συμφωνία ως προς το πόσο θα πρέπει να καθοριστούν οι νέοι ευρωβουλευτές αλλά το Συμβούλιο το 2008 είχε συμφωνήσει ότι ε, μπορούν ε, οι χώρες ή να συγκαλέσουν μερικές εκλογές ή να καθορίσουν ε, εκπροσώπους του Εθνικού Κοινοβουλίου και ίσως όλα αυτά δεν συνάδουν με τις διατάξεις και γι' αυτό προσπαθούμε να βρούμε μία λύση με τον συνάδελφο Μέντες Δεβίγκο. Αν όμως παρακολουθήσουμε τη συζήτηση στη Γαλλία, από ό,τι κατάλαβα, ο Πρωθυπουργό ζήτησε από τον πρόεδρο της Βουλής να ε, καθορίσει ε, δύο ε, εκπροσώπους από το ΕΛΚ πράγμα που οφείλεται σε ένα λανθασμένο και περίπτωση περίπλοκο σύστημα στη Γαλλία. Μέχρι στιγμής όμως δεν θα μπορέσουν να καθοριστούν οι δύο αυτοί μέχρι το τέλος του χρόνου. Δηλαδή δεν θα μπορέσουν να έρθουν καν μέχρι το τέλος του 2010. Έτσι εγώ αντιλαμβάνομαι την κατάσταση. Εάν θέλουμε λοιπόν να εξηγήσουμε σαφώς την κατάσταση για τους πολίτες μας θα πρέπει να κάνουμε κάτι γρήγορα και αποτελεσματικά διότι η συνέλευση κρατάει πολύ χρόνο. Μπορούμε να να την επιλέξουμε, μπορούμε όμως να κάνουμε και άλλες επιλογές, να ξέρουμε τι κάνουμε, αλλά ό,τι και να κάνουμε πρέπει να είναι σαφές και απλό και αποτελεσματικό για τους πολίτες. Δεν βλέπω άλλους να ζητούν το λόγο και έτσι ο κύριος Νταφ τώρα ε, ζήτησε ε, άπαξ και άκουσε τις απόψεις ο κύριος Φερβέρ όμως εκπρόσωπος του Συμβουλίου μήπως θέλει να σχολιάσει. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Νόμιζα ότι είχαμε την ευτυχία και την ευλογία να παρίσταται ένας εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πράγμα όμως το οποίο φαίνεται δεν ισχύει και αν δεν είναι δεν μπορεί να μιλήσει. Εφόσον λοιπόν θα συνεχίσει η συζήτηση στα θέματα αυτά ε, τα συνταγματικά, καλό θα ήταν να μας ε, στείλει το Συμβούλιο έναν εκπρόσωπο που θα μπορέσει να λάβει το λόγο επί του θέματος. Ποιος ζήτησε ακόμη να μιλήσει? Ο Γκουαλτιέρη. Δεν θα ήθελα να καταχραστώ τις ε, επίοικιά σας θα ήθελα να μόνο σε κάτι που είπε η Γαλλίδα συνάδελφος. Κάτι δεν καταλαβαίνω. Υπάρχει ένα επιχείρημα που λέει επιλογή ότι αν γίνει επιλογή εκτός της Βουλής θα υπάρξουν προσφυγές. Οι βουλευτές ορίζονται από τα κράτη έτσι και αλλιώ με οποιαδήποτε λύση, αφού οι εκλογέ έχουν γίνει. Επομένω, δεν μπορεί να γίνει προσφυγή κόντρα εναντίον μιας απόφασης της ε, Βουλής στη συγκεκριμένη περίπτωση που θα όριζε του δύο βουλευτέ. Οι, προ... οι λύσει 2 και τρία είναι διαφορετικέ. Δηλαδή, η δυνατότητα, οι δυνατότητε είναι δύο. Ή θα έχουν εκλεγεί από τους πολίτες με νέες εκλογές ή θα οριστούν από την κυβέρνηση από το κράτος. Πρώτη υποϋπόθεση, αν υπόψη τα αποτελέσματα των τελευταίων ευρωεκλογών. Δεύτερη υποπερίπτωση, από βουλευτές. Αλλά ουσιαστικά αυτός που ορίζει το βουλευτή δεν είναι υπογείτες. είναι το κράτος. Προσφυγή λοιπόν κατά της επαφασιβής δεν έχει νόημα. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, αυτό μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι αυτή η πρόταση τροπολογίας του Συμβουλίου δεν είναι απόλυτα σαφής, γιατί ουσιαστικά φαίνεται να είναι τρεις λύσεις, ενώ δεν είναι τρεις λύσεις σε ίδια βάση και οι τρεις συνταγματικά. Αυτή τη διευκρίνηση μόνο έπρεπε να κάνω, έκρινε σκόπιμο να κάνω. Μέντες Δεβίγκο, για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρο. Το πρώτο σχόλιο που ήθελα να κάνω είναι για να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους συμμετείχαν με πολύ ενδιαφέρουσες ε, παρεμβάσεις όπως πάντα σε αυτή την Επιτροπή με επιχειρήματα που θα εμπλουτίσουν όχι μόνο τη συζήτηση όπως τα έκανα αλλά και το κείμενό μου. Πρώτα απ' όλα, συμφωνώ με τον κύριο Νταφ. Καλό θα ήταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η Προεδρία, κάποιο εν πάση περιπτώσει, να είναι παρόν και να μπορέσει να λάβει το λόγο ή να μας πει ποια είναι η θέση του Συμβουλίου. Πρέπει να ψηφίσουμε. Καλό θα ήταν. Επίσης, θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι από αυτά τα οποία είπε και η κυρία Γιαννάκου και ο κύριος Σόλτ και ο κύριος Φόξ σε σχέση με τους τρεις Γερμανούς βουλευτές. Δεν είναι θέμα λήψης απόφασης κατομοφωνία για να εγκαταλείψουν τη θητεία τους ενδεχομένω οι τρεις συνάδελφοι. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αδύνατο. Έχουν εκλεγεί και δεν μπορεί να υπάρξει εκ των υστέρων απόφαση που να το στείλει σπίτι τους. Και αυτό είναι ίσως κάτι το οποίο δυσχεραίνει την κατάσταση, αλλά εν πάση ζούμε σε, σε ε, κοινωνίες δικαίου. Δεν υπάρχει θέμα για αυτούς τους τρεις συναδέλφους. Και νομίζω ότι το θέμα αυτό είναι σαφές να μην χάσουμε χρόνο. Εξελέγησαν για πέντε χρόνια και θα συνεχίσουν ως το τέλος της θητείας του Παρόντος Κοινοβουλίου. Ας μην τριγυρίζουμε γύρω γύρω γύρω γύρω από αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει δυνατότητα να αλλάξει μια τέτοια ηλυμένη απόφαση. Δεύτερον, πιστεύω ότι κανένας από τους παρεμβαίνοντες δεν είπε ότι είναι αντίθετος με τη σύγκληση μιας διακυβερνητικής. Και αυτό μας ερωτά το Συμβούλιο. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριοι, είστε υπέρ του να συγκληθεί διακυβερνητική για το θέμα αυτό. Άρα, εφόσον κανεί δεν είναι αντίθετο, συμφωνούμε. Κάποιοι είπαν ότι θέλουν, προτιμούν convention, συνέλευση. Άλλο αυτό. Αλλά, καταρχήν, η ιδέα τη σύγκληση μια διακυβερνητική για να επιληθεί ένα πολιτικό θέμα, μια πολιτική απόφαση έτσι όπως ελήφθηκε, εξήγησε ο κύριο Χάουρεγγι, είναι κάτι το δεδομένο. Είχαμε μια πολύπλοκη κατάσταση, όπως ξέρουμε, πριν από την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας που πέρασε από διάφορα εμπόδια και υφάλους, αλλά είχε ληφθεί μία πολιτική απόφαση άλλαξαν τα πράγματα με τη θέση σε ισχύ. Όπως ξέρετε πέρασε μια εκτενέστατη περίοδος ε, επικύρωσης της νέας επιτροπής. Ξέρετε πολλές φορές περνάνε μήνες ολόκληρους. Βάσει περιπτώσει τα πράγματα δεν εξελίσσονται πάντα όπως τα είχαμε προβλέψει. Άρα έχουμε ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο εδώ πρέπει να λύσουμε. Τώρα, η συμπερίληψη των 18 βουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημαίνει ότι σεβόμαστε μία πολιτική απόφαση που είχαν λάβει οι αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων και έχουν κυρώσει όλες οι βουλές. Άρα πρόκειται για μία πολιτική συμφωνία. Θα έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 751 και όχι 735 βουλευτές. Πράγμα που σημαίνει ότι σχεδόν για όλες τις χώρες μας θα υπάρχουν ισορροπίες ισορροπίες ε, που θα γίνουν και κατά την λήψη αποφάσεων στο Συμβούλιο και για μας. Έχουμε περιπτώσει κρατών που έχουν λίγους βουλευτές και το να έχουν περισσότερους σημαίνει ότι εκπροσωπούνται καλύτερα στα πλαίσια της, ε, του πλουραλισμού αν θέλετε που είναι το πνεύμα που μας διέπει εδώ και θα λύσουν και κάποια εσωτερικά προβλήματα στους κάθε χρόνος. 12, 12 χώρες αφορώνται από το θέμα αυτό, δεν είναι λίγε. Λοιπόν, και εδώ συμφωνούμε, κανένας δεν εξέφρασε αποκλίνουσα άποψη. Τώρα, Φυσικό είναι να υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις για τον τρόπο με τον οποίο θα ενεργήσει το Συμβούλιο. Όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι εγώ δεν ξέρω πώς θα το πούνε οι διερμηνείς. Ε, για κάτι το οποίο έγινε και δεν έγινε όπως θέλαμε, αλλά έγινε με κάποιο τρόπο, εγώ δεν κλαίω. Ό,τι έγινε, έγινε. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να επανέλθουμε. Είχαμε ειδοποιήσει όμως ότι θα γίνουν έτσι τα πράγματα και είχαμε προειδοποιήσει και το Συμβούλιο. Προσέξτε πώς πρέπει να ενεργήσετε. Όπως πάντα. Και σε αυτή την περίπτωση. Δεν άκουσε τι λέμε. Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, όχι το, το, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Έπρεπε, είπαμε, πέρσι το Μάρτιο με τσεχική προεδρία να έχει πάρει μία σχετική απόφαση. Μας περιπτώσει. Ξέρουμε τι συνέβη σε αυτή την ατυχή ε, τσεχική προεδρία. Δεν το είχε και ω προτεραιότητα το θέμα αυτό. Έπεσε η κυβέρνηση στη μέση του θητεία του, είχαν άλλα προβλήματα. Το Εν πάση περιπτώσει, Εν πάση περιπτώσει, αν είχε ληφθεί μια τέτοια απόφαση, δεν θα είχαμε το πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε τώρα. Αλλά τώρα, εφόσον προέκυψε, Πρέπει, αντί να κλαίμε για το τι έγινε πέρσι, να λύσουμε το πρόβλημα τώρα. Το Συμβούλιο, λοιπόν, που έχει λάβει την καταρχήν πολιτική απόφαση, τι μας ζητά. Να ανοίξει ο δρόμος για να μπορέσει κατά κάποιο τρόπο να επιληθεί το θέμα της προσχώρησης αυτών των 18 βουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα. Και Ξέρουμε για αυτό το θέμα πόσο, ε, τι πρόβλημα αντιμετωπίζει μία μία συγκεκριμένη χώρα. Η Γαλλία. Και θέλω να ευχαριστήσω την νέα συνάδελφο που στην ε, πρώτη της παρέμβαση χρειάστηκε να σχολιάσει την κατάσταση, τι που δεν είναι εύκολη. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι έχουμε δύο δυνατότητε πολιτικέ για να επιληθεί το θέμα αυτό. Η πρώτη έγκυται στο εξή. Α προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση και η άλλη είναι δεν θα δεχθούμε να έρθουν εδώ βουλευτές που δεν έχουν εκλεγεί άμεσα. Έχουμε αυτές τις δύο δυνατότητες. Από πολιτικής πλευράς και οι δύο απόψεις είναι υπερασπίσιμες. Αλλά ας μην κρυφτούμε πίσω από τη σύγκληση συνέλευσης ή ας μην προφασιστούμε κάτι άλλο για να μην λύσουμε το πρόβλημα ο καθένας σας παρουσιάσει τα ε, επιχειρήματά του. Και εγώ είμαι στη θέση σας. Εάν πει η πλειοψηφία της Επιτροπής μας, ποτέ δεν θα δεχθούμε βουλευτές να έρθουν, εάν δεν έχουν εκλεγεί με άμεση καθολική ψηφοφορία τον Ιούνιο, θα συμφωνήσω. Ας προσπαθήσουμε να υπερασπίσουμε αυτή την άποψη και δούμε τι θα γίνει. Αλλά μην κρυφτούμε πίσω από μια μάσκα που να λέει συνέλευση και που θα μας επέτρεψε να έρθουμε αντιμέτωποι με το Συμβούλιο και να αποκρύψουμε κατά κάποιο τρόπο την έλλειψη πολιτικής βούλησης. Ειλικρινά, πιστεύω ότι, και το λέω αυτό στον κύριο Φρεγόστορ με μεγάλη αγάπη, εγώ θαυμάζω τι έγινε στο Λάκελα το 97 εμείς την εφήβραμε αυτή την περίφημη κομβόσια. Εμείς. Και στην κολονία κάναμε τον χάρτη θεμελιωδών θυματών και πιστεύω ότι αυτή η convention, η συνέλευση ήταν πολύ μεγάλη ανακάλυψη. Πολύ πολύτιμη. Αλλά θα πρέπει να τη χρησιμοποιούμε όταν πρέπει να τη χρησιμοποιούμε. Επίσης, όπως λέμε στην Ισπανία, δεν χρειάζεται να βάλουμε κανόνι για να σκοτώσει μια μύγα. Δηλαδή, τι κάνουμε τώρα. Βάζουμε άλλο ένα στις δυνάμεις για να λύσουμε ένα μικρό πρόβλημα. Πιστεύω ότι πολύ δύσκολα θα πείσουμε την κοινή γνώμη ότι επειδή δεν μπορέσαμε έγκαιρα να λύσουμε το θέμα των δύο Γάλλων Ευρωβουλευτών, θα, θα συγκλίνουμε, θα, συγγνώμη, θα, θα επικαλεστούμε τη σύγκληση μια νέα συνέλευση για να δούμε πώς θα μπορέσουμε διαδικαστικά να αφήσουμε το... θέμα. Ακούστε, δεν είναι θέμα της παρούσης. Στο σημείο 5 του ψηφίσματος Ενδέχεται ενδεχομένως στο μέλλον να γίνει κάτι τέτοιο. Όταν υπάρχει σοβαρό λόγο. Ενδεχομένω. Εάν προσχωρήσει η Κροατία και κάτι πρέπει να κάνουμε για του Κροάτες συναδέλφου. Τότε ενδεχομένω θα μπορούσαμε να συγκαλέσουμε μια συνέλευση. Διότι αν τη συγκαλέσουμε τώρα για να λύσει ένα τόσο μικρό πρόβλημα και συγκεκριμένο, νομίζω ότι θα είναι σαν να υποτιμούμε τον ρόλο τον οποίο πρέπει να διαδραματίζει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω του συναδέλφου για τα σχόλιά του. πάση περιπτώσει, πιστεύω κύριε Πρόεδρε, και σήμερα πρέπει να σας πω ότι ολογνωμικά σας λέω και παροιμίως ε, από τη χώρα μου. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι ούτως ή άλλως κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσα να πω ότι ο κύβο έχει ρηφθεί, δηλαδή ξέρουμε περίπου τι πρέπει να κάνουμε και θα πρέπει να βρούμε την καλύτερη, την κατάλληλη λύση. Πιστεύω όμως ότι περαιτέρω συζήτηση δεν χρειάζεται να κάνουμε. Και όπως σας είπα, όπως και ο κύριος Νταφ, παρακαλώ, α είναι ένα εκπρόσωπος της ε, ε, Ισπανικής Προεδρίας εδώ για να συζητήσουμε μαζί του, διότι ξέρουμε ότι το Συμβούλιο έστειλε την επιστολή αυτή, ζητώντας να απαντήσουμε σε κάποια ερωτήματα. είναι λοιπόν κάποιος από το Συμβούλιο παρόν για να κάνουμε και μαζί του συζήτηση. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλες παραμονές. Δεν βλέπω άλλο να ζητάει το λόγο. Προτείνω λοιπόν να εγκρίνουμε την πρόταση του εισηγητή, να ορίσουμε ημερομηνία για τις τροπολογίες. Αν συμφωνείτε, προτείνω το εξή. Η ημερομηνία τροπολογίε. 11 Μαρτίου, 12 ώρα το μεσημέρι, ψηφοφορία 7 Απριλίου. Αν δεν έχουμε αντίρρηση, αποφασίζεται αυτό και περνάμε στο επόμενο σημείο, πολύ σημαντικό. Θεσμικέ πτυχέ προσχώρηση Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πράσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Η Νάφο Χαουρέγη μας έχει δώσει ήδη την έκθεσή του. Έχουμε και την γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελευθεριών με βάση το άρθρο 50 του κανονισμού. Ο συνάδελφος Χαουρέγγι ήδη μας έχει δώσει το κείμενό του. Έχει οριστεί ακρόαση για τις 18 του μηνός όλη την ημέρα, πρωί-απόγευμα, Νομίζω έχει μοιραστεί ο κατάλογος αυτών που θα έρθουν στην ακρόαση να μας μιλήσουν. Σχεδόν όλοι, με εξαίρεση έναν, είπαν ότι θα έρθουν, από, είναι από κάμποσα κράτη. Πρόκειται για επιφανείς προσωπικότητες Δεν χρειάζεται νομίζω να υποβάλουμε τροπολογίες πριν την ακρόση. Ας ακούσουμε τις υπερογνώμονες πρώτα. Δεν ξέρω αν ο εισηγητής, ο συνάφος ε, Χαορέγκοη, θα ήθελε να μας μιλήσει για το θέμα αυτό. Θέλει. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, διότι ήδη το είχα κάνει στην προηγούμενη συνάντησή μας. Απλώς θα ήθελα να επιβεβαιώσω, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος, ότι προβλέπουμε μία ακρόαση με την παρουσία εμπειρογνωμόνων και προσωπικότητων, την οποία θα οργανώσουμε στις 18 Τρίτου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα, δεδομένου ότι το θέμα μας έχει πάρα πολύ σημαντικές τεχνικές πτυχές. Λάβαμε υπόψη και διάφορες υποδείξεις που μας έκαναν οι άλλοι συνάδελφοι της Επιτροπής και πιστεύω ότι η ακρόαση της 18ης Τρίτου είναι πάρα πολύ σημαντική. Σε σχέση τώρα με την έκθεση που έχετε για τις θεσμικές προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση την πρόσφαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και λαμβάνοντας την ε, ε επί της ε, ουσίας έκθεση της Επιτροπής ΑΦΚΟ θα πω το εξή και την γνωμοδότηση τη ΕΒΕΣ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω, να υπενθυμίσουμε μάλλον το εξή. Με την προσχώρηση Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των πρόσφυγη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και την κύρωση του χάρτη των θεμελιωδών ελευθεριών που ενσωματώθηκε στη συνθήκη, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ή μάλλον η πολίτες της Ευρώπης, όλος ιδιαιτέρως μάλλον, προσχωρούν σε ένα πλήρες νομικό σύστημα το οποίο ζητούσε επί χρόνια η νομολογία και όλη η πολιτική κουλτούρα που μας διέπει. Δηλαδή να έχουμε ένα σύστημα τι το οποίο όλα τα δικαιώματα του ανθρώπου και όλα το κοινοτικό δίκαιο θα ενσωματώνονταν για να μπορέσει να υπάρχει μια σαφής άποψη επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτός και είναι ένας από τους στόχους προσχώρηση. Προσχώρηση, εξάλλου, δίδει μια νέα διάσταση προστασίας στα θεμελιώδη δικαιώματα σε παγκόσμιο επίπεδο και συμπληρώνει την εσωτερική προάσπιση αυτών των δικαιωμάτων από το δικαστήριο. Τι λέει η έκθεση. Όπως μπορέσατε να δείτε, σε 12-13 σημεία συνοπτικά λέει τα εξή η έκθεση. Πρώτα απ' όλα, περιγράφουμε τα επιχειρήματα υπέρ της προσχώρησης Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση, ε, επιπτώσεις της προχώρησης σε αυτό το νομικό σύστημα και κυρίως την παράγραφο 4 του πρώτου σημείου μιλούμε για τη σχέση μεταξύ δικαστηρίου ευρωπαϊκού και δικαστηρίου για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Στη δεύτερη παράγραφο τι λέμε. Αυτό το οποίο λέει συνθήκη. Η προσχώρηση δεν μπορεί να σημαίνει διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι συγκεκριμένη, πρόκειται για συγκεκριμένη εντολή που προβλέπεται και αναφέρεται στο σημείο το σχετικό της συνδίκης. Κατά την άποψή μου είναι ιδιαίτερα, σημαντικέ είναι ιδιαίτερα σημαντικές οι παράγραφοι 3 και 4, στις οποίες επίσης λαμβάνοντας υπόψη ποια είναι η εντολή της συνθήκης Λισαβόνας λέγει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σεβαστεί την ιδιαίτερη κατάσταση που ισχύει στα κράτη-μέλη σε σχέση με τη συνθήκη αυτή. Για κάθε χώρα χωριστά, έτσι όπως ισχύει σε κάθε χώρα. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι είναι σημαντικό να ξέρουμε βάσει ποιου πρωτοκόλλου, ποια συμφωνίε και με ποιο τρόπο γίνεται η προσχώρηση Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ευρωπαϊκή αυτή σύμβαση. Και αν αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω των πρωτοκόλων τα οποία έγιναν αποδεκτά ομόφωνα από τα κράτη-μέλη. Και συγκεκριμένα το 1, 2, το 4 και το 7. Στο σημείο 5. Λέμε ποιες είναι οι επιπτώσεις από αυτή την προσχώρηση, δηλαδή με ποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμμετέχει στα εκτελεστικά όργανα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, τη Μουλή τη Ευρώπη και πώς μπορεί να συμμετέχει στην εκλογή των δικαστών. Στο σημείο 6 αναφέρεται κατά κάποιο τρόπο η απαγόρευση προσφυγής ενός κράτου προς άλλο, δεν έχει νόημα κάτι τέτοιο και βεβαίως εφόσον όλα αυτά τα κράτη-μέλη είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπεται να υπάρχει τέτοια δυνατότητα ε, για τα κράτη-μέλη. Επίσης, ε, νομιμότητα των μέσων. Ποιος μπορεί να προσφύγει κατά ποιου. Ενεργός και παθητική προσφυγή. Αν πρόκειται για πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προσφυγή θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν πρόκειται για κάτι που αφορά ένα κράτο, κατά του κράτους. Και αν πρόκειται για κράτο μέλος και Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή το σύνορο, το ορόσημο μεταξύ των δύο είναι κάπως ασαφές, προβλέπετε πώς θα γίνεται. Επίσης, προβλέπετε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη μπορούν να, να είναι και οι δύο αντικείμενο προσφυγής. Δηλαδή, όποια και να είναι η αρχή κατά της οποίας προσφεύγει κάποιος, είτε είναι Ευρωπαϊκή Ένωση ή κράτος μέλος, μπορούν ως ανεξάρτητες οντότητες να ζητήσουν κάποιος να υπερψηφίσει τα δικαιώματά τους. Επίσης γίνεται λόγος σε επόμενες ε, παραγράφους για την προσφυγή που μπορεί να γίνει και τον διάλογο για να επιληθούν τα προβλήματα. Στην επόμενη παράγραφο λέγεται ότι το δικαστήριο θα πρέπει να είναι η πηγή έμπνευσης για την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο σημείο 11 γίνεται λόγος για την αναφορά το φόρτο, ο φόρτος εργασίας του Ευρωπαϊκού ε, δικαστηρίου να μπορέσει να αμφλυνθεί. όπως ξέρετε υπάρχει μεγάλο φόρτος εργασίας του Δικαστηρίου. και να μπορέσουν, διότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με μία επικύρωση εκκρεμή ακόμη από τη Δούμα της Ρωσίας, ώστε να μπορέσει να υπάρχει ε, απάλυνση του φόρτου εργασίας. Και στο σημείο 12 και τελειώνω, λέγεται ποια είναι η διαδικασία προσχώρησης. Και για να πω τα πράγματα πιο απλά, θα πω το εξής. Εδώ υπάρχουν πέντε βήματα τα οποία πρέπει να θυμόμαστε. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει εντολή διαπραγμάτευσης για την προσχώρηση, δηλαδή το Συμβούλιο δίνει εντολή στην Επιτροπή να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση. Δεύτερον, η διαπραγμάτευση, η ίδια διαπραγμάτευση για την ίδια τη διαπραγμάτευση. Δεύτερον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα πρέπει να εγκρίνει την πράξη προσχώρησης. Τέταρτον, αναφέρεται ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει ομόφωνα και στο πέμπτο και τελευταίο σημείο, το πέμπτο βήμα, το τελευταίο όλη αυτή τη διαδικασία είναι ότι θα πρέπει να γίνει η επικύρωση εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε προοδευτικά αυτά τα πέντε βήματα για να έχουμε την πλήρη προσχώρηση και αυτό είναι κάτι το οποίο θα τραβήξει χρόνο, αν θέλετε. Τελικά γίνεται αναφορά στο εξή η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την πρόσφυση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών μπορεί να αποτελέσει ενδεχομένως ένα πρώτο βήμα πριν να περάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσχώρησή της στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Επίσης, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να φερθώ σε μια απόφαση που έλαβε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 8 Φεβρουαρίου. Πρώτα απ' όλα, στην έκθεση του Συμβουλίου λέγεται, αναφέρονται κυρίως τα θέματα αυτά τα οποία προανέφερα. Αλλά για να ξέρετε, πώς διαμορφώθηκε η πολιτική τους επιχειρηματολογία, θα πω το εξή λέει, τα τέσσερα εξή σημαντικά του Συμβουλίου. Λέει το Συμβουλίο, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δούμε ποια είναι η εμβέλεια και το περιεχόμενο της προσχώρησης στην ε, σύμβαση και όπως είπα και προηγουμένως, θα πρέπει να πούμε σε ποια και σε πόσα πρωτόκολλα αναφέρεται αυτή η προσχόληση. Εγώ σας ανέφερα ότι αυτά τα πρωτόκολλα αναφέρονται σε σημεία 3 και 4 της εκθεσής μου. Δεύτερον, δεύτερο θέμα το οποίο έθεσε το Συμβούλιο. Η κατάσταση των κρατών μελών μετά από από την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ αναφέρεται ότι δεν μπορεί να γίνει διεύρυνση αρμοδιοτήτων. Λέγεται πώς θα γίνει η εξασφάλιση, η διασφάλιση το ότι κάθε κράτος μέλος κρατά τα δικαιώματα τα οποία είχε προσχωρώντας και δεν θα αλλάξει τίποτα με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης και βεβαίως αναφέρεται και το ε, δικαίωμα ερμηνεία του συνθήκη στην οποία έχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Επίσης, τι λέει στο τέλος το Συμβούλιο. Ότι πάντα, εάν υπάρχει προσφυγή, θα μπορεί να γίνει προσφυγή κατά ενός κράτους μέλους και κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εάν τεθεί κάποιο τέτοιο πρόβλημα, αν τεθεί πρόβλημα προσφύγη κατά τη Ένωση κράτους μέλου. Και τελευταία αναφέρεται η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εκπροσώπησή της στα όργανα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Πράγμα το οποίο σας είπα ότι συμπεριλαμβάνεται στο σημείο 5 της εκθεσής μου. Τελειώνει το Συμβούλιο και τελειώνω κι εγώ, λέει ο κ. Χουάργη, με δύο ερωτήματα τα οποία έθεσε στα κράτη-μέλη το Συμβούλιο. Εάν συμφωνούν, πρώτα απ' όλα να εγκριθεί η εντολή διαπραγμάτευσης για να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις ε, πριν από τον Ιούνιο. Πρώτα απ' όλα, διότι δεν τίθεται θέμα πρέπει να αρχίσει ή όχι η διαπραγματεύση. Αυτό είναι κάτι το οποίο προβλέπεται. Το ερώτημα είναι, συμφωνεί το Συμβούλιο να αρχίσουν οι δια... Ε, συγγνώμη, συμφωνεί το Κοινοβούλιο να αρχίσει το Συμβούλιο της διαπραγματεύσεις πριν από τον Ιούλιο. Διόνιο. Και δεύτερον, ερωτά κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει και μας ως Κοινοβούλιο. Ποιος θα είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Καταλαβαίνω ότι το Συμβούλιο εκφράζεται υπέρ της στενής σχέσης μόνιμης ενημέρωσης της Επιτροπής μας αυτό επιθυμεί περισσότερο το Συμβούλιο, αντί να θέλει κάποιο μέρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμμετάσχει απευθείας στην διαπραγματευτική ομάδα. Αυτά περιλαμβάνονται στην εκθεσή μου και, όπως σας λέγω, είναι θέματα τα οποία συζητώνται από το Συμβούλιο. Και βεβαίως, η πρόθεσή μας είναι να συνεχίσουμε να ακούμε τι έχει να πει το Συμβούλιο ε, σας λέγω και λυπάμαι που δεν το προηγουμένως, εγώ μίλησα με την κυρία Γιαννάκου που είναι εκπρόσωπος του ΕΛΚ για το θέμα αυτή και υπεύθυνη ώστε να μπορέσει η έκθεση αυτή να είναι μια έκθεση στην οποία θα συμφωνήσουμε όλοι μεταξύ μα. Έχω έρθει και θα έρθω και σε διαφορά και συζήτηση με τι άλλε ομάδε. Αυτό όμω το οποίο είναι σημαντικό είναι να γίνει η ακρόαση, μάλλον προβλέπεται στι 18, και εκείνη την ημερομηνία, εκείνη την ημέρα κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να εγκρίνουμε και ποια θα είναι και η καταληκτική ημερομηνία κατάθεση τροπολογιών και αφού συμφωνήσουμε με τις άλλες επιτροπές να καταλήξουμε και στην τελική ψήφιση έκθεση έκθεσης αυτής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει ο συνάδελφος Πρέντα, εισηγητής για γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που με υποδεχτήκατε στην επιτροπή σας και μου δώσετε το λόγο. Έκανα την γνωμοδότηση αυτή, αλλά δεν θα σας την παρουσιάσω με λεπτομέρειες, όπως έκανε ο εισηγητής σας. Θα ήθελα μόνο να υπογραμμίσω μερικά σημεία. Καταρχήν σας θυμίζω το ότι η συνθήκη της Λισαβόνας γενικά αναφέρει σε ενισχυμένη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην Ένωση και εκτός Ένωσης στη σχέση της με τρίτα κράτη και υπηκόους. Και ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι νομικά δεσμευτικός και το άρθρο 6, παραγραφός 2, ορίζει ότι η Ένωση υπογράφει την Ευρωπαϊκή Συνθήκη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Θεμελιώδεις Ελευθερίες και γι' αυτό στο σχέδιο γνωματοτησής μου υπογραμμίζω τρία βασικά σημεία. Το πρώτο είναι ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις τρίτε χώρες. Το δεύτερο, διαδικασία για την επιμερισμό αρμοδιοτήτων στην Ένωση. Και το τρίτο, η συμμετοχή με αντιπροσωπεία της Ένωσης στα διάφορα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το πρώτο σημείο. Διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις τρίτες χώρες το υπάρχει ένα χώρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο ισχύσει τον διάλογο αυτό με τους γειτονές μας προς Ανατολάς που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Συνθήκης Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και τότε θα έχουμε τις ίδιες υποχρεώσεις. Εμείς ως Ένωση. Και αυτή θα βοηθήσει γενικά στην αύξηση και του κύρους της Ένωσης έναν των τρίτων χωρών. Δεύτερον, διαδικασία. Το πρωτόκολλο 8 της Συνθήκης Λισαβόνας προβλέπει να οριστεί ένας μηχανισμός για επιμερισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης. Όταν υπάρχουν όμως αμφιβολίες, θα πρέπει να οριστεί ποιος είναι ο κάθε εταίρος με βάση τη συνθήκη υπό τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Και τρίτο, η συμμετοχή μέσω αντιπροσωπείας της Ένωσης στα διάφορα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Όπως είπε και ο κύριος Χουαλέγγι στην έκθεσή του, η Ένωση θα πρέπει το δικαίωμα να συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου στι συνεδριάσει του Υπουργικού Οργάνου, σε ορισμένε περιπτώσει, όταν ασκεί το ε, ελεγκτικό ρόλο τη ή όταν γνωμοδοτεί, προκειμένου να ζητηθεί γνωμοδότηση από το δικαστήριο και να εκπροσωπείται στην Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που όπως ξέρετε είναι όργανο της ε, Υπουργικής Επιτροπής. Εγώ στη δική μου έκθεση υπογραμμίζω την ανάγκη δημοκρατικού ελέγχου εκ μέρους του Κοινοβουλίου στη διαδικασία ορισμού του εκπροσώπου ή των εκπροσώπων της Ένωσης στην Υπουργική Επιτροπή και της Διευθυντικής Επιτροπής όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, Κομιτέ Directeur. Τέλος, στη γνωμοδότησή μου επισημαίνω το δικαίωμα το Ευρωκοινοβούλιο να ορίσει, να αποστείλει εκπροσώπους στην ε, κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης όταν συζητιόνται συναφή θέματα. Θα πρέπει να φροντίσουμε η αρμόδια επιτροπή στο Κοινοβούλιο να εκπροσωπείται στην ειδική αυτή αντιπροσωπεία. Θα βάλω και επιπλέον πληροφορίες με βάση αυτά που είπε ο εισηγητής σας πιο πριν. Η ψηφορία τον Ιανουάριο ο σε επικύρωση του πρωτοκόλλου 14 της συνθήκης και θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει από την 1η Ιουνίου. Γιατί έχει κλείσει ήδη ο κύκλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε και εμείς. Ήλκια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επειδή προηγουμένως δεν μίλησα, θα ήθελα τώρα να μιλήσω ε, και να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά που έκανε και για τον ε, τρόπο με τον οποίο συγκέντρωσε όλα τα στοιχεία και ε, που τα παρουσίασε εις ε, την Επιτροπή Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Όσον αφορά το σχέδιο της εκθέσεως και του ψηφίσματος, δεν μπορούμε να πούμε ότι όλα έχουν απαντηθεί, ήταν ε, προφανές και πιστεύουμε ότι αυτά τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη εύκολα μπορούν να, ε, να υιοθετηθούν κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε ε, στα ερωτήματα που ακόμη κυκλοφορούν. Δηλαδή, τις διαφορές μεταξύ των αρμοδιοτήτων των δύο ε, δικαστηρίων, του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου και του Δικαστηρίου του Στρασβούργου. Το ένα Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το άλλο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πιστεύω ότι το θέμα αυτό θέλει περισσότερη προσοχή και περισσότερη επεξεργασία διότι όταν μιλάμε για τις αρμοδιότητες των δύο δικαστηρίων ε, μιλάμε για θέματα τα οποία ίσως ε, γνωρίζουν οι δικαστικές αρχές αλλά που δεν είναι θέματα που μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν για να ξεκινήσει μία αναδιοργάνωση. Δεύτερον, η αναμόρφωση ε, του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είχε προβλεφθεί στη, στα σχόλια την προηγούμενη φορά. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η αναμόρφωση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν θα αναδιαρθωθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ώστε να υπάρχει μία διασύνδεση ε, διότι διαφορετικά η δομή ε, το, του ο, Δικαστηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα θα είναι πάρα πολύ περίπλοκη, ήδη είναι πολύ περίπλοκη και ε, θα υπάρξουν από τη συγχώνευση πιο πολλά προβλήματα παρά λύσεις δεν νομίζω ότι τα κοινοτικά δικαστήρια θα σταματήσουν να λειτουργούν. Θα καταφέρουν ίσως να λειτουργήσουν και με μεγαλύτερη ταχύτητα. Αλλά υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου η δυσαρέσκεια ορισμένων που απευθύνονται στα ευρωπαϊκά δικαστήρια θα γίνει αισθητή και ενδέχεται ε, ανταυτού να απευθυνθούν στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Άρα μία διαρθρωτική ε, συγχώνευση μπορεί ήδη να εξετάζεται κατά τρόπον ώστε ε, όλα τα δικαστήρια ε, να μπορούν να λειτουργούν σε όλα τα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως πιο συγχρονισμένα. Και τέλος, γνωρίζουμε ότι όταν οι αποφάσεις του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρονται σε διάφορα θέματα των εθνικών νομικών συστημάτων μπορεί να οδηγήσουν σε τροποποίηση, αυτών των εθνικών συστημάτων ποια θα είναι τα αποτελέσματα για την Ένωση σε περίπτωση που η Ένωση ε, καταδικαστεί ε, ή τιμωρηθεί ε, από το δικαστήριο όταν θα έχει κυρωθεί το, το, η συνθήκη. Είναι, είναι θέματα που ίσως θα έπρεπε να εξετάσουν οι επιτροπές κατά τρόπον ώστε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα τα οποία θα είναι η εποδός αυτής της διαδικασίας. Όπως βλέπετε τα προβλήματα είναι πάντοτε πολύ ε, περίπλοκα και γι' αυτό ο, μου δίνετε το δικαίωμα να παρέμβω εδώ και να πω ότι η σχέση μεταξύ της ε, ενσωματώσεως ε, του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, είναι ε, κάτι το οποίο είναι προφανές αλλά όταν πρέπει κανείς ε, να συμφωνήσει ε, στις αποφάσεις του ε, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, των διαφόρων δικαστηρίων, ποια προέχουν και ποια ακολουθούν, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να εξετάσουμε στα πλαίσια της συνθήκης της γιατί είναι πολύ σημαντικό και πρέπει όλα αυτά να τα εξετάσουμε και να λάβουμε υπόψη ε, στην έκθεση η οποία θα καταρτιστεί. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Μπαφ. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ περίπλοκο. Και καλό θα ήταν η μετάφραση από τα ισπανικά να είναι καλή σε όλες τις γλώσσες, το οποίο λυπούμε αλλά ε, δεν συντρέχει στην περίπτωση. Διότι εδώ πρέπει να ξέρουμε τι εξετάζουμε και τι δεν ε, συζητάμε. Ε, εάν δεν έχουμε εξαιρετική μετάφραση αυτό δεν επιτυχάνεται. Επίσης πρέπει να αιτιολογήσουμε την απόφαση να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε ε, εις ε, το, να έχουμε πρόσβαση στο Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με καλύτερο τρόπο από ό,τι τώρα. Δηλαδή, η σημασία των αποφάσεων από τους συντάκτες της συνθήκης για πρόσβαση εις το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας επαναφέρει στο θέμα ε, της συνθήκης η οποία ήταν μια συμβιβαστική λύση για να μπορέσει η χάρτα να γίνει δεσμευτική και γι' αυτό συμφωνήσαμε να μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση η ε, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ήταν ε, ε, μία συμβιβαστική λύση μεταξύ των Βρετανών οι οποίοι απεχθάνονταν την ιδέα του συνταγματικού χάρτη και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο ήθελε να υπάρχει ένας ε, προεξέχων κατάλογος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών αρχών. Οπότε όλα τα θέματα αυτά μπορούν να γίνουν κατανοητά από μας και από τα εθνικά πολιτικά κόμματά μας και τους δικαστές. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μπορούμε να εξηγήσουμε σε αυτή την έκθεση ε, και δεν θα το εξηγήσει βέβαια το Συμβούλιο θα πρέπει η πρόσβαση στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να συμπληρώσει την απόφαση ο χάρτης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να καταστεί υποχρεωτικά, υποχρεωτικός και ε, θα βοηθήσει στην εφαρμογή του χάρτη πλήρως και αποτελεσματικά όσον αφορά τις αρμοδιότητες τις οποίες έχουμε αποκτήσει ε, στα θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν είναι σωστό όπως λέγεται στην παράγραφο 2 ότι η προσχώρηση ε, δεν ε, συνεπιφέρει μία επέκταση των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως διότι δεν νομίζω ότι δεν είναι σωστό ότι δεν υπάρχει κάποια επέκταση. Ίσως, ίσως αυτό ευθύνεται, γι, αυτό, γι' αυτή τη διατύπωση ευθύνεται η αγγλική μετάφραση. Δεν ξέρω αν τα ίδια λέγονται ισπανικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν συμφωνώ. Και εφόσον ε, θα υπάρχουν δικαστές του δικαστηρίου στο Στρασβούργο θα υπάρχει μία επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και εφόσον μιλάμε για αρμοδιότητες πιστεύω ότι η πρόσβαση στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν συνεπιφέρει ε, διεύρυνση αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά πρέπει να διαχωρίζουμε τις εξουσίες των θεσμικών οργάνων από τις άλλες. Όσον αφορά την παράγραφο 5, πολύ σωστά ο εισηγητής λέγει ότι υπάρχουν τρία πράγματα τα οποία επακολουθούν τις αποφάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μπορούμε δηλαδή να διαβεβαιώσουμε ε, ότι έχουμε δικαίωμα να προτείνουμε τρεις υποψηφίους. και να τους επιβάλλουμε στην Επιτροπή των Υπουργών αλλά θα πρέπει να υπάρξει μία διαδικασία για την ερμηνεία αυτών των δικαιωμάτων για να μπορέσουν να εφαρμοστούν, για να μπορεί ε, να αιτιολογηθεί μία εσωτερική απόφαση που θα αναφέρεται στην επιλογή των υποψηφίων φαντάζομαι ότι η εντολή της Επιτροπής η οποία θα μας εκπροσωπήσει στην ε, Επιτροπή των Υπουργών θα είναι αυτή. Άρα ε, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χαρουέγγι για αυτό αλλά νομίζω ότι ακόμη έχουμε δρόμο μπροστά μας προτού μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ε, τα ερμηνεύουμε σωστά. Η κυρία Γιαννάκου έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή με τον οποίο έχουμε κάνει ήδη συζήτηση όπως ο ίδιος είπε για την έκθεση αυτή. Πραγματικά ενώ φαίνεται ε, ότι είναι μία απλή υπόθεση προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην ουσία ανακύπτουν πάρα πολλά ζητήματα και πάρα πολλά ερωτήματα. Καταρχήν ε, θεωρητικός η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων προστατεύει εξίσου με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όμως οι μέχρι σήμερα αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έχουν κατά κάποιο τρόπο δημιουργήσει δεδικασμένο και υπάρχει δια της προσχώρησης αυτής ευρύτατη κατά κάποιο τρόπο προστασία που μπορεί ίσως, ίσως σε αυτό το σημείο ο κύριος Ντάφνα έχει δίκιο, να επιφέρει και διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης. Όχι άμεση, έμεση όμως, λόγω των μέχρι σήμερα αποφάσεων. Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα σημεία πάντως, ε, σε κάθε περίπτωση είναι ε, ο διεθνής χαρακτήρας προστασίας που είναι πολύ σημαντικός και είναι και σημαντικός ε, για ε, τα πρόσωπα από τις τρίτες χώρες. Είναι σημαντική η ανάγκη του θεσμικού συντονισμού των δύο ευρωπαϊκών δικαστηρίων, ο οποίος επιτυγχάνεται βέβαια με την προσχώρηση της Ένωσης στην Σύμβαση των Δικαιωμάτων και την υπαγωγή συνακόλουθα στον έλεγχο της σύμβασης αυτής με τη συμβατότητα του κοινοτικού δικαίου. Βεβαίως εδώ ανακύπτουν ερωτήματα σε σχέση με τις χώρες που δεν έχουν αποδεχθεί την εφαρμογή της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο εδαφός τους, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, ενώ ταυτόχρονα έχουν κυρώσει τη Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ε, ποιας εφαρμογής δηλαδή και ποια προστασία την χάνουν τα άτομα ε, στις χώρες αυτές. Φυσικά στα ευρωπαϊκά κράτη η βασική προστασία προέρχεται από τη συνταγματική τάξη του κάθε κράτους Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουμε όλο και περισσότερες υποθέσεις και περισσότερα ζητήματα τα οποία τελικά ε, επιλύονται μέσω του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ιδιαίτερα ζητήματα που αφορούν σε αποζημιώσεις παραδείγματο χάρη ε, στη χώρα μου κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80 έγιναν από το Σοσιαλιστικό Κόμμα πάρα πολλές κρατικοποιήσεις διαφόρων επιχειρήσεων ε, Εν συνεχεία σε ερώτηση που έκανα ως εθνικός βουλευτής τι έχει γίνει με αυτό το θέμα, απεκαλύφθη ότι η Ελλάδα πλήρωνε εξωφρενικά ποσά αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες των κρατικοποιημένων επιχειρήσεων διότι δεν είχε τηρήσει ε, μια συγκεκριμένη ε, τάξη δικαιωμάτων η οποία προβλεπόταν από τη Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επομένως, είναι, ε, η υπόθεση δεν είναι πάρα πολύ απλή Υπάρχουν πολλές πλευρές. Παραδείγματο χάρη αν μπορούν κάποιοι να προσφύγουν ένα κράτος μέλος εναντίον της Ένωσης, η Ένωση εναντίον ενός κράτους μέλους, οι πολίτες αντιστοίχως και βέβαια ποιος θα καθορίζει το δικαστή που θα συμμετέχει στο, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, τέλος, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που νομίζω θα το συζητήσουμε με τον εισηγητή, στο άρθρο 13 αναφέρεται και στην ε, επιθυμία κατά κάποιο τρόπο της ε, Ένωσης να προσχωρήσει στον κοινωνικό χάρτη του 1961, όπως τροποποιήθηκε στο Στρασβούργο το 1996 και στον οποίο δεν έχουν προσχωρήσει περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι καταρχήν θέλω να συγχαρώ και πάλι τον εισηγητή. Είναι μεγάλο το βάρος που έχει πέσει στους ώμους του. Νομίζω ότι η ακρόαση που θα πραγματοποιήσουμε με τις ε, νομικές προσωπικότητες τις οποίες έχουμε καλέσει και που έχουν κατά καιρούς ασχοληθεί ιδιαίτερα με το ζήτημα αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ ε, και βεβαίως ε, θα μας εισαγάγει σε λεπτομέρειες οι οποίες καταρχήν δεν είναι εμφανείς αλλά μπορούν να γίνουν πάρα πολύ εμφανείς ε, εν συνεχεία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ το Συμβούλιο στις αποφάσεις αυτές αναλύοντας περισσότερο το ζήτημα αυτό και μπαίνοντας περισσότερο στο βάθος και μην κρατώντας ε, μόνο μια τυπική διαδικασία δεδομένου ότι εάν ε, ο τρόπος προσχώρησης δεν είναι σωστός τελικά μπορούν να παρουσιαστούν μεγάλα νομικά ζητήματα στο μέλλον και ανάμεσα στα κράτη-μέλη και ανάμεσα στα δύο δικαστήρια που και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Uh, <clears throat> Ευχαριστώ είναι ένα ερώτημα που έθεσα και προηγουμένως αλλά είχα αντιφατικές απαντήσεις και όταν ρώτησα την Ισπανική Προεδρία μου είπαν δεν ξέρω, περιμένετε και θα δούμε. Δηλαδή, όταν θα προσχωρήσουμε στην συνθήκη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα αποτελέσει νόμο ή θα είναι μία διεθνή σύμβαση την οποία έχουμε προσχωρήσει προσυπογράψει διότι εάν ε, αποτελέσει μέρος της νομοθεσίας του Ευρωπαϊκού ο, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν θα ισχύσει μόνο για το δικαστήριο του Στρασβούργου αλλά και του Λουξεμβούργου. Ε, με απλά λόγια. Ναι ή όχι. Έχω δίκιο ή όχι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θέλω να συγχωρώ τον κύριο Χάουρικη για την εξαιρετική δουλειά που έκανε. Βέβαια, το θέμα είναι εξαιρετικά προβληματικό. Πολύπλοκο. Πρόκειται για ένα θέμα για το οποίο όλοι συμφωνούμε. Ακόμη και ο τελευταίο ε, συνάδελφο φαίνεται να συμφωνεί ότι η προσχώρηση καλό πράγμα Αλλά τελικά έχουμε μία συμφωνία καταρχήν, αλλά βλέπουμε τώρα τι δυσκολίε διότι πρόκειται για ένα πολύπλοκο θέμα. Όταν είμαστε εκεί τότε και συντάσαμε και συζητούσαμε το χάρτη μελεδών δικαιωμάτων, το θυμάται κύριο Νταφ, είχαμε θέσει κάποια ερωτηματικά. Κάτι που θα ήθελα να συμμεληθεί είναι το εξή. Η προσχώρηση στην σύμβαση αποτελεί μέρος πολιτικής ε, συμφωνίας που συμπεριλαμβάνει τον υποχρεωτικό χαρακτήρα του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και πολλοί εκπρόσωποι τον μελών είπαν ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει πρόβλημα δεδομένου ότι έχουμε δύο διαφορετικές δικαιοδοτικές αρχές για αυτά τα θέματα στην Ευρώπη, όπως λέγεται. Αν θυμάστε, τότε με μία επιστολή την οποία είχαμε συντάξει, προσπαθήσαμε με τις τελικές διατάξεις να αποτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή, όταν στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων αναφέρεται κάτι το οποίο πηγάζει από τη συνθήκη της Ρώμης, εμείς στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίδαμε την ίδια έννοια που προσέδιδε και η συνθήκη της Ρώμης. Υποχρεωτικός λοιπόν χαρακτήρας του χαρτί έτσι όπως θα ε, συμπληρωθεί εκ των υστέρων. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό είναι αυτό το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην πρώτη παράγραφο που μιλάει για την αρχή της ανεξαρτησίας του κοινοτικού δικαίου. Το Στρασβούργο είναι εν τέλει υπεύθυνο και εγγυάται τελικά τα δικαιώματα τα οποία εξασφαλίζει η Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αλλά τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία εξασφαλίζουν και εγγυώνται αυτά τα δικαιώματα ο καθένας στη χώρα του. Δεν πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό δικαιοδοτικό όργανο που το κάνει αυτό εξ ονόματος όλων. Και τελικά Εάν κάποιο σε εθνικό επίπεδο δεν ικανοποιηθεί από κάποιες αποφάσεις, προσφεύγει στο Στρασβούργο, δεν υποκαθιστά το δικαστήριο του Στρασβούργου, κανένα εθνικό δικαστήριο. Έτσι θα συνεχίζουν να είναι τα πράγματα και πρέπει να είναι απόλυτα σαφές για όλους. Ένα άλλο σημείο το οποίο θα ήθελα να τονίσω και νομίζω ότι είναι σημαντικό, ότι στην πρώτη συζήτηση που είχαμε αυτό παρέμεινε κάπως εκρεμές και περιμέναμε να λυθεί κάποια απόφαση. Το σημείο 6 το αναφέρει και σωστά ο συνάδελφος. Το θέμα της διακρατικής προσφυγής μιλάμε για συνεργασία μεταξύ μας και ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να προσφύγουμε σε εξοκοινοτικό δικαστήριο να λύσουμε αν θέλετε ενδοκοινοτικό πρόβλημα. Αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό και πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους και είναι κάτι το οποίο είχαμε συζητήσει την πρώτη φορά αλλά ίσως ακόμη ήταν ε, όχι απόλυτα σαφέ για όλου. Στην Μαδρίτη, στα πλαίσια τη Προεδρία, οργανώθηκε ένα σεμινάριο. Ο Ατόνιο Βιτορίνο, που είναι καλό μα φίλο όλων, είπε κάτι το οποίο θέλω να αναφέρω εδώ. Ο... Τι τον απασχολεί στο Βιτορίνο. Πώς γίνεται η προσχώρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης στην σύμβαση και τι σημαίνει με τις εξαιρέσεις και τις επιφυλάξεις. Διότι έλεγε ότι θα μπορούσε να υπάρχει να υπάρχουν κάποια δικαιώματα τα οποία εξασφαλίζονται στην Ένωση και τα οποία θα μπορούσε κάποιος να μην μπορεί να εξασφαλίσει διότι εκφράζονται επιφυλάξεις. Θα πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα γιατί είναι σημαντικό. Επίσης, πιστεύω ότι θα πρέπει να αποφανθούμε για ένα άλλο θέμα το θέμα της εκπροσώπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμβούλιο Υπουργών όταν πρόκειται για μια περίπτωση στην οποία καταδικάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δεκαετία του 80 ήμουν μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, ήμουν από την άλλη μεριά αν θέλετε και θα πω πολλές φορές και το λέω ευγενικά ότι πολλές φορές τα κράτη εφήρμοζαν με πάρα πολύ με αργό τρόπο κάποιες αποφάσεις. Σπρώχναν κάποιοι, αλλά εκείνοι οι κύριοι παίρνουν τον χρόνο τους. Είναι λοιπόν σημαντικό να ξέρουμε στην συγκεκριμένη περίπτωση ποιο θα μας εκπροσωπήσει. Εάν ε, εκτιμήσει ότι υπάρχει κάποια παρέκκληση, παραβίαση το δικαστήριο, ποιος θα εκπροσωπήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το θέμα είναι ένα θέμα στο οποίο εγώ ακόμη δεν έχω απάντηση και νομίζω ότι καλό θα ήταν να το σκεφτούμε περαιτέρω, να το μελετήσουμε περαιτέρω. Και τελικά κύριε Πρόεδρε, υπάρχει κάτι άλλο θετικό που το λέει και σωστά η έκθεση. Στο σημείο 9. Όλοι θέλουν να έχουν κάποια βεβαιότητα όταν συζητούμε θέματα όπως η σύμβαση, η προσχώρηση, η σχέση μεταξύ του δικαστηρίου στο Λουξεμβούργο με το δικαστήριο Στρασβούργο, βλέπουμε ότι υπάρχει πειρασμός μεταξύ των υποθετικών προβλημάτων που ενδεχομένως θα μπορούσαν να παρουσιαστούν, να προσπαθούμε να βρούμε ένα μέσο διαφέτησης των προβλημάτων, έναν τρόπο να βρούμε λύσεις. Και αυτό τα λέει πάρα πολύ σωστά η εκθέση στο σημείο 9. Θέλουμε κάποια βεβαιότητα. Όλοι θέλουμε σε κάποια πράγματα να έχουμε βεβαιότητα ότι κάτι θα γίνει σωστά. Αλλά το δίκαιο δεν δίνονται πάντα βεβαιότητες για κάτι. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα παρθούν ε, οι σωστές λύσεις και θα βρεθούν οι σωστές λύσεις από το Λουξεμβούργο και, ή από το Στρασβούργο. Ναι, όπως προσπαθούν να κάνουν όλα τα δικαστήρια, ακόμη και τα συνταγματικά. Αλλά θα πρέπει εμείς να βρούμε έναν τρόπο να επιλύουμε τα προβλήματα, δεν ξέρω, ή μέσω μιας ε, ομάδας ε, ή μέσω μιας δικαθυσίας, σε πάση περιπτώσει, που θα μπορούσε να επιλύσει τον τρόπο. Είμαστε, ζούμε όλοι σε κράτη δικαίου, υπάρχουν προβλήματα, μπορούν να πετεθούν προβλήματα ερμηνείας, αλλά νομίζω ότι η υπερίσχυση ποιου σε σχέση με κάποιον άλλον είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι απόλυτα σαφές. Και τελευταίο σχόλιο, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σκεφτούμε ακόμη περισσότερο κάτι στο οποίο αναφέρθηκε και ο εισηγητής την εντολή διαπραγμάτευσης της Επιτροπής, πώς θα συμμετάσχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Ο πειρασμό θα είναι να μας αφήσουν ε, κατά μέρο. Και γι' αυτό μιλούν για στενή συνεργασία και στενή σχέση. Την ξέρουμε αυτή τη στενή σχέση. Εγώ θα ήθελα να πω το εξή. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να συνεισφέρει στην εξέβρεση λύσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να κάνει κάτι. Θα ήθελα λοιπόν να σκεφτούμε πώς θα μπορέσει να συνδεθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην διαπραγμάτευση. Διότι στα πλαίσια της ακρόασης που θα κάνουμε για να μελετήσουμε κάποια θέματα, νομίζω ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε πολύ περισσότερο από το να πούμε κάποια στιγμή της διαδικασίας «Ναι, συμφωνώ, όχι, δεν συμφωνώ». Ευχαριστώ κυρία, κύριε Γκοδεμέντες, κυρία Γκουρμάη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον συντονιστή για την εξαιρετική εργασία. Συμφωνώ με τον ε, συνάδελφο ότι πρόκειται για ένα πολύ περίπλοκο θέματα, θέμα, ε, ότι χρειάζονται διαβουλεύσεις και όταν το εξετάζω διαπιστώνω ότι πολλά από τα σημεία έχουν καλυφθεί. Άρα πάμε καλά στην έκθεση αυτή ε, έχουν ε, ε, έχουν παρατεθεί τα περισσότερα επιχειρήματα γιατί πρέπει να προσχωρήσουμε σε αυτή τη σύμβαση που είναι σημαντική για μας και θα πρέπει ε, συγχρόνως να ενισχύσουμε την συνταγματική σημασία μιας τέτοιας προσχωρήσεως σε αυτήν την σύμβαση και πιστεύω ότι ο εισηγητής έχει αναφέρει και τη δυνατότητα να υπάρξει μία ακρόαση, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υποχρεωμένο να έρθει σε επαφή με καλούς εμπειρογνώμονες και η Επίτροπος κυρία Ρέντινγκ προφανώς θα μας παρουσιάσει μία πολύ καλή επισκόπηση του θέματος. Θέλω να συγχαρώ λοιπόν και πάλι πάλι τον εισηγητή και είμαι βέβαιη ότι το έγγραφο στο οποίο θα καταλήξουμε θα είναι εξαιρετικό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα υπάρξουν ε, ταραχές εις ε, τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όταν θα προσυπογράψουμε αυτή τη ε, συνθήκη διότι το 1986 ήδη είχαμε εξετάσει, είχαμε πει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μέρος του κεκτημένου. Άρα υπήρχε πάντοτε ενδιαφέρον, αλλά προκύπτουν και προβλήματα και γι' αυτό πολύ σωστά έχουμε οργανώσει την ε, ε, ακρόαση πριν πάρουμε οποιαδήποτε απόφαση όταν θα γίνει αυτή η ακρόαση θα πρέπει να εξετάσουμε όλα τα θέματα που μπορούν να καταστήσουν πιο περίπλοκη αυτή τη διαδικασία. Δεν θέλω να κάνω μια πολιτική συζήτηση γιατί αυτό θα γίνει μετά την ακρόαση αλλά θέλω να επανέλθω σε ένα θέμα που ήδη θίξαμε δηλαδή μέχρι ποιου σημείου οι δικαστές πρέπει να συμμετέχουν όταν ένας από τους ε, δύο ε, ενδιαφερόμενους ε, είναι ένας διάδικος είναι της χώρας τους. Ε, είναι κάτι που θα πρέπει να εξεταστεί. Μας είχε λεχθεί ότι δεν είναι πρόβλημα διότι τότε ε, ο δικαστής αυτός θα απέχει από το να ε, εκδώσει ετοιμιγορία όταν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά υπάρχουν προβλήματα αρμοδιοτήτων για αυτούς τους δικαστές και θα πρέπει η έκθεση να εξετάσει και αυτό το σημείο. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να μπορέσουμε να επανεξετάσουμε αυτό το θέμα. Δεν θα δώσω συνέχεια, αλλά περιμένω τα αποτελέσματα. Ε, Πρωτού δώσω το λόγο στο συνάδελφο Χαραουή, θα ήθελα να αναφερθώ σε μεθοδολογικά θέματα σχετικά με την απόφαση. Πρώτον, φυσικά δεν μπορούμε να προτείνουμε τροπολογίες πριν, πριν γίνει η ακρόαση. Μάλλον μπορούμε να, να προτείνουμε είναι όμως μάλλον ανάγκη, επειδή το θέμα είναι περίπλοκο, να δώσουμε στον εαυτό μας λίγο χρόνο να σκεφτούμε το θέμα μετά την ακρόαση. Διότι, για να ικανοποιηθεί η Ισπανική Προεδρία να κλείσουν οι εργασίες αυτές, έτσι ώστε να δοθεί εντολή στην Κομισιόν μέσα στο πρώτο εξάμεινο, αμέσως μετά την ακρόαση θα έπρεπε να βάλουμε ημερομηνία για τις τροπολογίες. Θεωρείτε ότι αυτό είναι λογικό. Δεύτερο ερώτημα. Οι ακροάσεις είναι σημαντικές και από τη συζήτηση βλέπω ότι υπάρχουν υψηλές προσδοκίες ως προς τις ακροάσεις. Θα έπρεπε να ζητήσουμε από τους ε, εμπειρογνώμονες να μας πούνε τη γνώμη τους για το πολύπλοκο αυτό θέμα ερωτώ ή θα ήταν σκοπιμότερο ο εισηγητής και επιμέρους βουλευτές ή ο πρόεδρος να θέσουμε συγκεκριμένες ερωτήσεις πριν την ακρόαση για να μην χάνουμε χρόνο και ακούμε δύο και τρεις φορές τα ίδια πράγματα. Ο το λόγο. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι μου φαίνονται όλες οι παρεμβάσεις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους και τα λοιπά. Νομίζω ότι θα δώσω κάποιες απαντήσεις, αλλά θα μπορέσουμε ίσως να έχουμε και κάποιες απαντήσεις μετά την ακρόαση. Για να απαντήσω στον πρόεδρο θα πω το εξή. Πιστεύω ότι όλη η επιτροπή μας όντως θα ήθελε να έχει περισσότερο χρόνο για την κατάθεση των τροπολογιών. Προφανώς στις 18 οι πραγματογνώμονες θα απαντήσουν σε ερωτήσεις που θα υποβάλουν όλοι μας. Οι ερωτήσεις που έγιναν εδώ και πολλές άλλες που μπορούν να τεθούν θα αποτελέσουν μέρος του πυρήνα της συζήτησης που θα γίνει τότε και από όσο καταλαβαίνω δεν χρειάζεται εδώ να αναλάβω όλες τις τροπολογίες. Στον κύριο Μέσερμις ένας εθνικός δικαστής θα του πει ότι το θέμα το οποίο θέτει προβλέπεται από κάποιους κανόνες και προδιαγραφές κάποιου δικαστηρίου. Θα του το πει κάποιος δικαστής. Είναι λοιπόν λογικό ο συνάδελφος να θέσει το ερώτημα στον δικαστή καθώς και όλοι οι συνάδελφοι, ο κύριος Μπρόνς, οι άλλοι σε σχέση με το τι συμβαίνει με το εθνικό δίκαιο κάθε φορά και την προσχώρηση στην σύμβαση να απαντηθούν όλα αυτά από τους ειδικού. Λογικό είναι στην ακρόαση της 18 Μαρτίου να ακούσουμε τι έχουν να πούνε οι ειδικοί και μετά από 8-10 μέρες να ε, έχουμε χρόνο για να καταθέσουν τις τροπολογίες. Νομίζω ότι λογικό θα ήταν να έχουμε κανένα δύο εβδομάδες μετά την ακρόαση για να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε και ο καθένας να καταθέσει τις τροπολογίες που επιθυμεί να καταθέσει. Και από εκεί εγώ θα προσπαθήσω με τη δική σας συνδρομή να βρω ένα συνενετικό κείμενο, ένα κείμενο το οποίο θα ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα, στα μελήματα, στις επιθυμίες του καθενός Και βεβαίω, εγώ δεν λέω ότι πρόκειται για πρώτη στο ενδιαφέρον τη Ισπανική Προεδρία. Δηλαδή δεν θέλω οπωσδήποτε το θέμα αυτό να συζητηθεί επί τη ε, ισπανική ε, προεδρία. Εγώ φαντάζομαι ότι οι συζητήσει στο Συμβούλιο δεν θα γίνουν πριν από τα μέσα ε, Μαΐου και εμείς μέχρι τότε φαντάζομαι ότι θα μπορέσουμε να έχουμε εγκρίνει έκθεση αυτή στην Ολομέλη. Τώρα, αυτό όσον αφορά τη μεθοδολογία πάρα πολύ σύντομα όμως, διότι μάλλον θα μπορέσουμε όλα αυτά τα θέματα να τα ξανασυζητήσουμε, όπως είπαμε μετά 18. Και θέλω να επαναλάβω κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση με τον διαφορετικό ρόλο που διαδραματίζουν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Το Ευρωπαϊκό το Δικαστήριο είναι εξειδικευμένο. Υπάρχει το δίκαιο και το κάθε εθνικό δικαστήριο. Το κάθε εθνικό δικαστήριο επίσης, επίσης πρέπει να πω ότι ασχολείται με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέχρι στον υψηλότερο βαθμό του και στην Ευρώπη. Αυτός ο οποίος ε, Ε, είναι, αν θέλετε, το ίστατο δικαστήριο για την ε, σωστή εφαρμογή όλων αυτών των δικαιωμάτων και ό,τι αφορά το κοινοτικό δίκαιο είναι το δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Είναι αυτό το οποίο έχει, αν θέλετε, τον τελευταίο λόγο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, ε, μια, μια οργάνωση, αν ένας πολίτης θεωρεί ότι μετά από τα ανώτατα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαιοδοτικά όργανα κατά την άποψή του. Υπάρχει ακόμη ένα δικαίωμα τα οποία δεν γίνεται σωστά σεβαστό, μπορεί να προσφύγει στο Στρασβούργο. Έχει το δικαίωμα να το κάνει. Και εδώ εμφανίζεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που επαγρυπνεί για αυτά τα δικαιώματα και προστατεύει αυτά τα δικαιώματα έτσι όπως τα θεσπίζει η σύμβαση, στην οποία θα προσχωρήσουμε και είναι, όπως είπαμε, υποχρεωτικά. Γιατί αποτελούν μέρος του κοινοτικού δικαίου και η Ευρωπαϊκή Ένωση <coughs> πρέπει να τα αυτά τα δικαιώματα. Όλοι, όλοι υποβάλλονται λοιπόν σε αυτή την δικαιοδοτική ε, τάξη, αν θέλετε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί? Διότι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέλη του δικαστηρίου. Και γιατί θέλει να προσχωρήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό είναι μέλος του DNA της, αν θέλετε. Πώς να το πω. Ε, εάν λοιπόν μας χαρακτηρίζει όλους, είναι ότι όλοι είμαστε εμβαπτισμένοι στα ίδια δικαιώματα στις υποχρεώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν θέλετε. Έτσι έχουν τα πράγματα και ευτυχώς που τα πράγματα έχουν γίνει με συστηματικό τρόπο. Και με την συνθήκη της νίκης, που είναι μέρος της συνθήκης τώρα, της συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι ήδη αποτελεί μέρος της συνθήκης, άρα είναι υποχρεωτικό δικαίωμα, άρθρο 6, Τι ρόλο παίζει το δικαστήριο. Εξωτερικό όργανο που προστατεύει όλα αυτά τα δικαιώματα στα πλαίσια αυτής της σύμβασης. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να είναι απόλυτα σαφές για όλους. Προτείνει κάτι που μου φαίνεται ενδιαφέρον ο κύριο Νταφ. Να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες πολιτικές εξηγήσεις, να γίνει περισσότερο παιδαγωγικού περιεχομένου, θέλετε, η δική μας παρέμβαση. για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε καλύτερα κάποια πράγματα. Ο κύριο Ντάφ, ο κύριο Μέντε Δεβίγο που ήταν οι πρωταγωνιστές όλης αυτής της ε, ε, διαδικασία για την, ε, το Σύνταγμα τη Ευρώπη, αν θέλετε σωστά έκαναν τις απαιτήσεις που έκαναν και θα πρέπει να αναφέρουμε όντως αυτό το προστατευτικό πλαίσιο των δικαιωμάτων των πολιτών. Και αυτό, όπως λέγω, είναι κάτι που είναι μέσα στο DNA της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ σωστά, λοιπόν, είπε ότι θα μπορούσαμε να τα αναφέρουμε αυτό που λέτε. Η μόνη μου δικαιολογία είναι ότι δεν θέλησα εγώ να είναι εκτενέστατη η έκθεσή μου, διότι ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια όρια όσον αφορά τον αριθμό των λέξεων, των ε, ε, σελίδων σε μια τέτοιου είδους έκθεση. Εγώ όμως, αν θέλετε, πραγματικά είμαι υπέρ της υπόδειξης που κάνατε. Τώρα, η αναφορά στο θέμα των αρμοδιοτήτων. Ακούστε, εμείς τι κάνουμε. Στη συνθήκη προβλέπονται κάποιες ε, εντολές που έχουν δοθεί στον καθένα. Ξέρετε ότι είναι, ε, βάζουν πάντα φρένο τα κράτη-μέλη. Α, προσέξτε, αυτό δεν θέλουμε να αποτελέσει ε, αύξηση των αρμοδιότητων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς ξέρουμε ποιες είναι οι αρμοδιότητες μας, ξέρουμε ποια είναι τα δικαιώματά μας. Απλώς αυτό το οποίο κάνουμε εδώ είναι αναπαραγωγή, αναπαραγωγή του κειμένου που μας επιβάλλεται από τη συνθήκη. Δεν ξέρω αν υπάρχει πρόβλημα γλωσσικό στα αγγλικά. Τέλος πάντων. Τώρα, το θέμα της, ε, του ορισμού των δικαστών. Αν θέλετε μπορώ να καταθέσω τροπολογίες για αυτό το θέμα, αλλά είχα την εντύπωση ότι στην έκθεση θα πρέπει κυρίως να πούμε τι σημαίνει η προσχώρησή μας όσον αφορά την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, αν θέλουμε εδώ να μιλήσουμε για διαδικασία, για την πρόταση επιλογής των δικαστών, Ξέρω, θέλετε να το κάνετε, α, άμα έχετε τέτοιου είδους ιδέες, δεν ξέρω. Τώρα, αμφιβολίες. Ο κύριος Πρέντα, εκπρόσωπος της ε, ΑΦΕΤ, μας είπε ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την εκπροσώπηση Ευρωπαϊκής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κοινοβουλευτική συνέλευση. Αυτό είναι κάτι για το οποίο έχω κάποιες αμφιβολίες. Δεν θα γίνει εύκολα, δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα είμαστε παρόντες, έχει νόημα, διαρωτώμε. Δεν μας εκπροσωπούν εμάς τα 27 κράτη-μέλη παρόντα, τα, 27 μέλη παρόντα στη συνέλευση αυτή. Επίσης, Κύριοι συνάδελφοι, Συγγνώμη που μπήκα σε τέτοιε λεπτομέρειε όσον αφορά κάποιε διαδικασίε, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η συζήτηση για τον θέμα του ρόλου που μπορούμε να διαδραματίσουμε εμείς σε όλη αυτή τη διαδικασία ε, διαπραγμάτευσης. Θα ήθελα πω στου δύο συναδέλφους που έκαναν τις ερωτήσεις, τις συγκεκριμένε, ότι το ότι ο δικαστής κάποιας χώρας δεν ψηφίζει όταν πρόκειται για δική της χώρας του υπόθεση είναι κάτι το οποίο ε, υπόκειται σε κανόνες οι οποίοι ορίζονται από τους κανονισμούς των δικαστηρίων. Βέβαια είναι πάντα παρόν για να δώσει κάποιες πληροφορίες αλλά ε, δεδομένου ότι ο κάθε δικαστής ξέρει κάποια πράγματα για τη χώρα του αλλά δεν ψηφίζει, δεν ψηφίζει στην τελική ε, ψηφοφορία. Αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει στα δικαστήρια. Αυτά ήθελα να πω συνέλθει. Και ακούστε, στις 18 πιστεύω ότι θα κάνουμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά με την ακρόαση. Θα ακούσουμε τι έχουν να πούνε οι εμπειρογνώμονες. Ας έχουμε κανένα δύο εβδομάδες στη θέση μας για να καταθέσουμε τροπολογίες, για να καταλήξουμε σε τροπολογίες με τις οποίες θα μπορέσουμε όλοι να συμφωνήσουμε και να έχουμε ένα κείμενο στο οποίο θα συμφωνήσουμε. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ. Τελειώσαμε τη συζήτηση αυτή για να κάνουμε τα πράγματα σωστά θα πρέπει να το σκεφτούμε πρώτα. Προθεσμοί για τις τροπολογίες τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά την ακρόαση. Ας πούμε 25, 25 Μαρτίου. Τι λέτε. Όχι πριν τις 25 Μαρτίου. Τώρα. Αν θέλουμε να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα της Ισπανικής Προεδρίας και λοιπά να κλείσουμε στο πρώτο εξάμεινο Αν και το πρώτο για μας είναι να κάνουμε τα πράγματα σωστά, θα πρέπει να αντέξουμε στην πίεση να πάμε πολύ νωρίς στην Ολομέλεια ή αφού υποβληθούν οι τροπολογίες να ψηφιστεί στην Επιτροπή μας παρακαλώ ακούστε με επαναλαμβάνω αν θέλουμε να τηρηθεί η προθεσμία του εξαμήνου θα πρέπει να έχουμε μια έκτακτη συνεδρίαση. Αν αντίθετα θεωρείτε ότι δεν υπάρχει λόγος να κλείσουμε άρον-άρον το θέμα αυτό μέχρι το τέλος Ιουνίου, τότε η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα γίνει αργότερα. Μέντες. Πρόεδρε, εγώ πιστεύω ότι εδώ δεν έχουμε μία πρώτη έκθεση του Συμβουλίου που περιμένει για να αρχίσει τη διαπραγμάτευση Ευρωκένους. Νομίζω ότι όπως είπε και ο συνάδελφος κ. Χουάραγκη, ας έχουμε χρόνο να σκεφτούμε τι, ποιες τροπολογίες θα καταθέσουμε και πώς θα κάνουμε σωστά τα πράγματα. Και σε σχέση με τους προσκεκλημένους μας την ακρόαση. Δεν θα πρέπει να ορίσουμε την, κατα... την προθεσμία κατάσταση τροπολογιών αμέσω μετά την αύξηση. Θα πρέπει να έχουμε λίγο χρόνο να το σκεφτούμε. Η εντολή του Συμβουλίου για την διαπραγμάτευση δεν νομίζω ότι εξάρτηται από την έκδοσή μα. Δεν είναι απαραίτητη προπόθεση. Να, τον λάβουν κάποια στοιχεία υπόψη, ή καλώ, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε και ε, εκτακτέ συνεδριάσει. Το λέγω αυτό διότι δεν νομίζω ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ του μεν και του δε. Αλλά όντω επειδή υπάρχουν θέματα πολύπλοκα πρέπει να έχουμε χρόνο στη θέση να μελετήσουμε πάρα πολύ καλά το όλο πρόβλημα. Ας μην τρέχουμε λοιπόν, ας μην βιαζόμαστε, με ηρεμία και περίσκεψη ας αντιμετωπίσουμε το όλο θέμα. Ευχαριστώ. Η γραμματεία μας προτείνει 26 Μαρτίου, 25 Μαρτίου για τις τροπολογίες. Οπότε ψηφοφορία στις 4 Μαΐου και ολομέλεια 14 Ιουνίου. Πρέπει να έχουμε δείξουμε ευελιξία, μα κάθε φορά να κάθε να κρίνουμε. Κανονίσουμε την ταχύτητά μας καθοδόν. Προτείνω λοιπόν. 25 Μαρτίου τον Απρίλιο στην Ολομέλεια και τον ε, στην Επιτροπή μας και τον Ιούνιο στην Ολομέλεια. Τώρα το πρόβλημα είναι ότι φτάσαμε σε 6 ώρα και έχουμε ακόμα τουλάχιστον δύο θέματα αρκετά σημαντικά. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να είμαι όσο πιο σύντομη γίνεται στις παρεμβάσεις μας. Προσαρμογή του κανονισμού στη συνθήκη της Λισαβόνας. Συγητής David Μάρτιν. Σας θυμίζω ότι ήδη εγκρίθηκε μια πρώτη ομάδα τροπολογιών για τη δεύτερη ομάδα που δεν θεωρήθηκαν ότι συνδέονται στενά με τη συνθήκη της διαβάσης είναι μια πρώτη αναβολή 25 Νοεμβρίου και στις 8 Φεβρουαρίου νέα αναβολή για τις τροπολογίες αυτές. Είμαστε στο νεκρό σημείο. Ο τύπος των τροπολογιών που δεν εγκρίθηκαν είναι αυτές που αναφέρονται στις σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια, επιμερισμός ε, ευθυνών μεταξύ Προεδρίου και Ολομέλειας και οι ασυλίες. Η αιτιολόγηση όσον αφορά τις ασυλίες, η βουλευτική ασυλία. Ένα από τα θέματα με βάση τα οποία αποφασίζεται αυτό το stand-by, δηλαδή να μπουν στο ψυγείο προς το παρόν αυτές οι τροπολογίες, παρότι σε εγκρίναμε ως Επιτροπή, είναι το ότι ορίστηκε, ενιστήθη μια ομάδα εργασίας για τις σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια και τη συνεργασία αυτή. Το Μάιο θα καταθέσει την έκθεσή της αυτή η ομάδα. Έπειτα οι τροπολογίε που δεν εγκρίθηκαν μέχρι στιγμή δεν αναφέρονται όλες στη σχέση με τα εθνικά κοινοβούλια. Η μελέτη λοιπόν των προβλημάτων και των σχέσεων με τα εθνικά κοινοβούλια έχουν ιδιαίτερη σημασία φυσικά σε σχέση με τις τροπολογίες που προτείναμε, διότι εμείς μας απασχολεί μόνο η μέθοδος, η διαδικασία. Θα ακούσουμε βέβαια τον εισηγητή μας. Υπάρχουν όμως πολιτικές δυσκολίες. Μπορεί να τις ξεπεράσουμε μια συμφωνία μεταξύ μας ή αν αυτό δεν γίνεται, δεν ξέρω, θα δούμε. Θα δούμε καταρχήν να δούμε τι έχει να μας πει ο εισηγητής μας, ο κύριος Μάρτιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάνατε μία πολύ εκτενή εισαγωγή, οπότε θα είμαι σύντομος ε, έχετε δίκιο. Βρισκόμαστε σε μία ε, κατάσταση εκκρεμότητος διότι βλέπουμε ότι υπάρχουν θέματα τα οποία ακόμη είναι προσυζήτηση, κανείς δεν ενδιαφέρεται να τα συζητήσει. Υπάρχει μία δύσκολη διαδικαστική κατάσταση γιατί η έκθεση αυτή δεν παραπέμφθηκε στην Επιτροπή, απλούστατα προχώρησε στην Ολομέλεια, δεν ε, εκτελέστηκαν όλες οι ψηφοφορίες. Έχουμε δηλαδή όλε, όλα τα, όλες τροπολογίες. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε νέες προθεσμίες, ε, νέο χρονοδιάγραμμα, δεν μπορούμε να σταματήσουμε, αλλά όπως είπατε έχουν αλλάξει οι συνθήκες, διότι υπάρχουν ομάδες εργασίας ε, με τα εθνικά κοινοβούλια, ε, δεν πρέπει να προχωρήσουμε αν δεν διαβουλευτούμε με τα εθνικά κοινοβούλια κοινοβούλια, τα θέματα είναι πιο αμφιλεγόμενα, δηλαδή ε, προκύπτουν συνεχείς δυσκολίες και η μόνη, δυσκολία, η μόνη λύση την οποία μπορώ εγώ να προτείνω είναι είτε να ψηφίσουμε αυτές τις τροπολογίες του Ολομέλεια και να αφήσουμε στη σοφία του Κοινοβουλίου τα περαιτέρω ή να περιμένουμε ως το Μάιο. Αλλά ε, μας είχαν πει ότι θα συζητηθεί στην Ολομέλεια τον Ιανουάριο. Και το τρίτο είναι η Επιτροπή αυτή να υιοθετήσει ατύπως συμβιβαστικές λύσεις που μπορώ να προτείνω σαν εισηγητή. Ο εισηγητής μπορεί να προτείνει συμβιβαστικέ τροπολογίες αφού έχει κλείσει η περίοδος για την υποβολή τροπολογιών και τουλάχιστον κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει η Επιτροπή αυτή να εκφράσει μία σαφή γνώμη σχετικά με τα θέματα που εκκρεμούν ακόμη. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι η πρόταση του εισηγητή με ικανοποιεί και θα την ακολουθήσω. Δεν πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα αυτά ε, σε ένα κενό ε, κρεμότητα Πρέπει να τα επιλύσουμε και γι' αυτό δέχομαι την πρόταση την οποία έκανε ο κύριος Μάρτιν. Ευχαριστώ κύριος Νταφ. Και εγώ συμφωνώ. Υπάρχουν και ορισμένα άλλα θέματα τα οποία έχουμε διαπιστώσει από όταν ίσχυσε το... η συνθήκη. Δηλαδή δεν έχει κλείσει το θέμα μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα ευγενές συμβιβασμό στην Επιτροπή και μετά να το προωθήσουμε και να το περάσουμε και από την Ολομέλεια. Κύριε Μάρτιν, θέλετε να αντιδράσετε. Πολύ σύντομα. Ε, χαίρομαι που με στηρίζει ο κύριος Μάντες Δεβίγο και ο κύριος Νταφ. Το μόνο που θέλω να πω στον κύριο Νταφ είναι ότι ειλικρινά πρέπει να σας πω ότι ουσιαστικά θα είμαστε ε, στην, ε, στην κρίση των υπηρεσιών εάν ε, πρόκειται να δεχθούν νέες τροπολογίες διαφορετικά μπορούν να τις θεωρήσουν απαράδεκτες. Γι' αυτό μίλησα για ένα ευγενή συμβιβασμό, glorious compromise. Και εγώ χαίρομαι που όλα αυτά γίνονται με ομοφωνία και δεχόμαστε την πρόταση του κυρίου Μάρτιν, τον οποίον καλούμε ε, να εκπονήσει τροπολογίες διάφορες και θα μπορέσουν να παρουσιαστούν στην συνεδρίασή μας της 17ης Μαρτίου. Με συγχωρείτε. Έχουμε 17 και 18 συνεδρίες, 18 έχουμε την ακρόαση, άρα ε, τροπολογίες για τις 17. Και πάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Είναι τέσσερις, ε, τέσσερα θέματα προς κοινή συζήτηση ε, που έχει αναλάβει ο κύριος Μέντες Ντεβίγκο που αναφέρεται στην εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και του ότι ε, προκάλεσε οικονομική κρίση. Φυσικά οι θεσμικές πτυχές, διότι η αρμόδια επιτροπή είναι η οικονομική επιτροπή. Εμείς μόνο θα γνωμοδοτήσουμε τρεις για τις ε, υποπτικές αρχές όσον αφορά την τράπεζα, Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, μία για τις κινητές αξίες και αγορές και το άλλο ασφαλείς και επαγγελματικές συντάξεις και για τη σύσταση μιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή Συμβουλίου για το συστημικό κίνδυνο, αποτροπής των κινδύνων. Ο κύριος Μέντες Δεβίγκο έχει το λόγο. Eh, Θα προσπαθήσω, κύριε Πρόεδρε, να κάνω πάρα πολύ συνοπτική παρουσίαση, βοηθούμενος από το PowerPoint. Πριν να μπω στα τεχνικά θέματα και, τον τροπολ... και στις τροπολογίες που αφορούν αυτές τις τέσσερις εκθέσεις να πω το εξής. Το 2008 η κρίση των χρηματοπιστωτικών μέσων και των αγορών έκανε τους Ευρωπαίους να ξυπνήσουν και να δουν ότι το ρυθμιστικό σύστημα ήταν ανεπαρκές και το ότι δεν υπήρχε επίσης σωστό σύστημα εποπτείας του όλου συστήματος. Αυτή η κρίση λοιπόν οδήγησε στο να γίνει μία μελέτη και το Σεπτέμβριο του 2009, ένα χρόνο μετά, η Κομισιόν δημοσίευσε τα αποτελέσματα ειδικής μελέτης, τα αποτελέσματα της μελέτης αν θέλετε. Αυτή είναι η πρώτη μου πολιτική αξιολόγηση. Λέγω ότι οι προτάσεις επιτροπέ είναι το μίνιμου μινιμόρουν τη πρόταση Λαβουασιέρ. Η Επιτροπή λοιπόν βλέποντα τι μπορεί να επιτύχει στο Συμβούλιο δεν ε, αντέγραψε κατά κάποιο τρόπο τις προτάσεις Λαβουασιέρ για τις παρουσιάσεις, τις έκανε κάπως πιο light, πιο ντεκαφεϊνέ θα έλεγα. Έτσι λοιπόν, αυτή η διαδικασία αποκορύφωσης αν θέλετε κατέληξε στο να μας δώσει αυτές τις προτάσεις ε, τόσο χαμηλού επίπεδου αν θέλετε. Και αυτό ίσως είναι πάντα ένα παιχνίδι που γίνεται. Έτσι λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι πολιτικό όργανο τώρα πρέπει να κάνει κάποιες πολιτικές κρίσεις. Εγώ θα σας παρουσιάσω το θέμα αυτό λέγοντας ότι επί της ουσίας είναι για την ε, άλλες επιτροπές μία κοινή δήλωση που είπαν θα θέλανε σε σχέση με τις προτάσεις Λαβουασιέ να πάνε πιο μακριά και από τις προτάσεις του Συμβουλίου και από τις προτάσεις της Επιτροπής. Εγώ προσπάθησα λοιπόν σε συνεργασία με τους εισηγητές της Επιτροπής ΕΚΟΝ να συνεργαστώ και πρέπει να πω ότι τρεις από αυτούς είναι από τους τέσσερις σχεδόν στην ίδια γραμμή πλεύσεως. Εδώ μιλούμε για τροπολογίες τεσσάρων προτάσεων της Επιτροπής. Και χρειάστηκε τη δουλειά να την ορίσουμε σε τέσσερα διαφορετικά θέματα, αν θέλετε. Πρώτα απ' όλα θα αναφερθούμε στις ε, συγκεκριμένες τροπολογίες που αφορούν την πρόταση της Κομισιόν και θα ήθελα τώρα να πω κύριε Πρόεδρε, σε υποφεληθούμε από τις οθόνες τις οποίες εμφανίζονται οι προτάσεις μας. Τι έχουμε. Πρώτα απ' όλα, το ευρωπαϊκό ε, νέο σύστημα εποπτείας, χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Είτε πρόκειται για τις ασφάλειες, είτε πρόκειται για τις τράπεζες, είτε πρόκειται για οτιδήποτε άλλο, για τις ε, συντάξεις, έχουμε να κάνουμε με εθνικές ε, ε, αρχές εποπτείας. Τώρα, το νέο σύστημα που προτείνουμε είναι όλα αυτά να γίνουν αντιστοίχως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και επίσης να συσταθεί και ένα νέο σύστημα, ένα νέο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το Συστημικό Κίνδυνο. Τι προτείνει αυτό το σύστημα. Διάφορα πράγματα. Εγώ τα παρουσιάζω συνοπτικά. Πρώτα απ' όλα, να θεσπίσει τεχνικές προδιαγραφές να εφαρμόζει με συνεκτικό τρόπο το κοινοτικό δίκαιο. Να παρεμβαίνει σε περίπτωση κατεπούσας ανάγκης. Να κάνει διευθέτηση των διαφορών. Να μπορεί να κάνει διευθέτηση των διαφορών διασυνοριακά όταν έχουμε να κάνουμε με δύο διαφορετικές οντότητες που είναι σε δύο ομορές χώρες και τελικά να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό ε, ταμείο ε, χρηματοπιστωτικής προστασίας αν θέλετε. Τώρα, ποιες θα είναι οι τεχνικές προδιαγραφές. Τι λέγει η πρόταση Επιτροπής. Η πρόταση Επιτροπής που είναι του Σεπτεμβρίου 2009 αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές είναι πράξεις που ανατίθενται βάσει των διατάξεων 209 της συνθήκης. Λέμε λοιπόν το εξής. Όταν θα πρέπει, αν υπάρχει μια ευρωπαϊκή αρχή διευθέτησης κάποιων προβλημάτων, εγκρίνει κάποιες διατάξεις αφού τις εγκρίνουν οι πάντες. Τι λέγει εδώ η πρόταση της Επιτροπής, ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή στέλνει αυτές τις προτάσεις στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πρέπει να τις εγκρίνει. Τι λέμε εμείς, τις στέλνει στην Εκομισιό και συγχρόνως τις στέλνει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Γιατί, δεδομένου ότι πρόκειται για αρμοδιότητες που ανατίθενται σε κάποιον. Τι γίνεται τώρα σε αυτή, με αυτό τον τεχνικό κανόνα που στέλνει ε, το σχέδιο στην Κομισιόν. Το εγκρίνει η Κομισιόν, το εγκρίνουμε εμεί, το εγκρίνει το Συμβούλιο, έχει καλώ. Τι συμβαίνει εάν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο δεν συμφωνήσουν με αυτέ τι προτάσει τη Κομισιόν. Τι μπορούν να κάνουν. Να πούνε και να κοινοποιήσουν ότι είναι αντίθετοι. Άρα δεν εγκρίνονται. Τι γίνεται τώρα εάν η Κομισιό δεν συμφωνήσει με ε, αυτή την την τεχνικό κανόνα τον οποίο θέλει να υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Αρχή. Δεν μπορεί να το κάνει. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως πρέπει να εγκρίνει και τι προσθέτουμε εμεί, ότι σε αυτή την περίπτωση το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερωθεί και το Συμβούλιο θα πρέπει να ενημερωθεί για του λόγου του οποίου την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Αρχή Επιτήρηση δεν την εγκρίνει η Κομισιόν. Εμεί θέλουμε περισσότερη Ευρώπη και βεβαίω περισσότερη διαφάνεια. Να μα λέει λοιπόν η Επιτροπή να έρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για να μα εξηγήσει γιατί απορρίπτει την πρόταση την οποία έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Αρχή Εποπτείας. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλω να πω είναι ότι αυτά τα οποία λέγω εγώ δεν υπάρχουν στην πρώτη επιτροπή. Επίση στην πρώτη επιτροπή δεν υπάρχει δυνατότητα που έχουμε να κάνουμε ανάκληση της, ε, του ε, δικαιώματος αυτού που έχουμε δώσει ε, ή της ανάθεσης μάλλον, ανάκληση της ανάθεσης. Όλα αυτά τα θέματα υπάρχουν στις εκθέσεις της Επιτροπής ΕΚΟΝ, με μια εξαίρεση, διότι μας λέγουν Μα λέει η ΕΚΟΝ ότι σε περίπτωση που υπάρχει κάποια διαφορά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερωθεί και η Επιτροπή Οικονομικών Υποθεσεων. Εμεί πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ενημερωθεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Και εγώ πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να μπούμε σε λεπτομέρειε, να πούμε ότι θα πρέπει να ενημερώνεται μόνο η Ευρωπαϊκή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Και συμφωνούμε με τι προτάσεις που υπάρχουν σε αυτές. Τώρα, κάτι άλλο το οποίο είναι επίση σημαντικό είναι συνεκτική εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Τι γίνεται αν μία εθνική αρχή δεν εφαρμόζει σωστά το κοινοτικό δίκαιο. Τι λέμε. Ότι αν γίνει προσφυγή εκ μέρους κάποιου αν δεν γίνεται σωστά η εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, δεν μπορεί να κάνει προσφυγή μόνο η Επιτροπή, αλλά το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο ή κάποιοι άλλοι. Και εδώ αναφέρονται οι δικές μας απόψεις, δηλαδή ε, ποια είναι η διαδικασία και ποιος μπορεί να κάνει μια τέτοιου είδους προσφυγή σε περίπτωση μη σωστής εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου. Τι γίνεται όταν υπάρχει κίνδυνος χρηματοπιστωτικής αστάθειας και πρέπει να γίνει κάποια ε, επίγουσα παρέμβαση. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό το οποίο λέμε είναι όχι μόνο η αρχή, η Ευρωπαϊκή Αρχή Εποπτείας σε περίπτωση επίγουσας ανάγκη να ζητήσει στο Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου να παρέμβει, αλλά να μπορεί και το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάμε λίγο παραπάνω λοιπόν από την πρόταση της Κομισιόν και λέμε, εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου θελήσει να παρέμβει, θα πρέπει να μας ενημερώσει και μας. Δηλαδή, ούτως ή άλλως, Πάντα θέλουμε να έχουμε ενημέρωση, πάντα να υπάρχει ενημέρωση των δύο υπευθύνων οργάνων για θέματα προπολογισμού, Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα, τι γίνεται σε περίπτωση επίσης που υπάρχει κάποια διαφορά, πώς γίνεται η διευθέτηση των διαφορών. Μιλούμε εμείς για την δυνατότητα διαμεσολάβησης Ευρωπαϊκής Αρχής Εποπτείας και αυτό το οποίο κάναμε, αυτό το οποίο προσθέσαμε εμείς είναι κάποιες διευκρινήσεις όσον αφορά τις προθεσμίες και ο καθορισμός κάποιων ε, πιο λογικών προθεσμιών από αυτές τις οποίες προέβλεπε η Κομισιόν. Και επίσης είπαμε ότι είναι αναγκαίο σε περίπτωση στην οποία υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των διαφόρων εθνικών αρχών εποπτείας σε σχέση με την ε, διαμεσολάβηση ή με τη συμφιλίωση που θέλουμε να γίνει η Ευρωπαϊκή Αρχή να μπορεί να λάβει μία υποχρεωτική, μία δεσμευτική απόφαση. Αυτό πιστεύω νομίζω ότι είναι λογική απόρρεια του συστήματος που θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα εποπτείας το οποίο να μπορεί κανείς μόνο προαιρετικά να λέει κάτι. Δεν πρέπει να έχει μόνο συστάσεις. Η αποφάση που λαμβάνει πιστεύω ότι σωστά θα πρέπει να είναι δεσμευτικέ. Εάν θέλουμε να εγκρίνουμε ένα τέτοιο σύστημα, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο σύστημα και αν θέλουμε περισσότερη Ευρώπη, θα πρέπει να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή αυτή αρχή εποπτείας ε, το δεσμευτικό αυτό χαρακτήρα. Τώρα υπάρχει κάτι καινούριο. Τι γίνεται σε περίπτωση που έχουμε διαφορές ε, διασυνοριακές μεταξύ εθνικών αρχών είναι κάτι το οποίο δεν προβλέπεται στην πρόταση της Κομισιόν. Το εισήγαγαν οι τέσσερι εισηγητέ τη επιτροπή ΕΚΟΝ και πάλι η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή είπαμε ότι παίζει διαμεσολαβητικό ρόλο και οι αποφάσεις της πρέπει να εφαρμόζονται από τις εθνικές αρχές. Αυτό είπαμε, είναι αυτό που θέλουμε, περισσότερη Ευρώπη. Και τελευταίο, μένα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων, των εξουσιών τους και της αποστολής τους είναι η και αφορά αυτό μόνο της, ε, το τραπεζικό σύστημα. Την σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστητικής Προστασίας που θα χρηματοδοτείται από τις συνεισφορές των χρηματοπιστωτικών και ε, ιδρυμάτων. Πρόκειται για ένα θέμα καινούριο, πρόκειται για ένα θέμα το οποίο θα προκαλέσει πάρα πολλές συζητήσεις γιατί είναι κάτι το νεοτεριστικό, αλλά όπως ξέρετε υπάρχουν ε, σε κάποιες χώρες για να προβληθούν τέτοιου είδους καταστάσεις κάποια εθνικά ταμεία εγγύσεων. Εμείς θα θέλαμε να γίνει κάτι τέτοιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι μου φαίνεται ότι σήμερα σε μια αγορά παγκοσμιοποιημένη, αλλά σε μια αγορά στην οποία δεν υπάρχει κανενός, κανενός είδους σύνορο, ε, το να περιορίζονται ε, κάποιες αρμοδιότητες σε εθνικό επίπεδο, ενώ οι τράπεζες ενεργούν χωρίς σύνορα, δεν είναι λογικό γι' αυτό. Θελήσαμε να εισαγάγουμε αυτήν την ιδέα τη δημιουργία αυτού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προστασία. Χωρί λοιπόν να θέσω ένα αμφιβόλο την ε, σε, ε, αρμοδιότητες και τη δυνατότητα των εθνικών συστημάτων να αντιδράσουν, η δημιουργία ενός τέτοιου Ευρωπαϊκού Ταμείου πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ λογική. Διότι θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να βρούμε σε περίπτωση τέτοιου είδους προβλημάτων ένα ευρωπαϊκό εποπτικό όργανο για να εφαρμόζονται κάποιες αποφάσεις οι οποίες θα πρέπει να ισχύουν για όλους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να πω ότι όλα αυτά τα θέματα, τα πολύ δύσκολα, τα πολύ πολύπλοκα, ε, μπορέσαμε με την ε, ε, Κλέρ να τα επεξεργαστούμε. Σας παρουσιάσαμε και σε γλώσσα που δεν είναι η δική μας γλώσσα συνοπτικά αυτές τις προτάσεις, τις οποίες κάνουν εξονόματος της Επιτροπή μας και επιμένω ότι οι προτάσεις αυτές έχουν γίνει στην ίδια γραμμή πλεύσεως με αυτό το οποίο κάνουν οι υπεύθυνοι επί της ουσίας. Συνεργάστηκα μαζί τους ώστε να μπορέσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να συμπεριλάβουμε τις δικές μας ιδέες και θέλω να πω ότι σε αυτό το στίχημα το μεγάλο των συναδέλφων της ΕΚΟ να κάνουν, ε, να ασχοληθούν με ένα τόσο σημαντικό θέμα για την Ευρώπη. Τη στιγμή την οποία όλοι θέλουμε περισσότερη Ευρώπη και τη στιγμή την οποία είδαμε ότι στα πλαίσια αυτής της οικονομικής κρίσης που μαστίζει όλους θέλουμε περισσότερη Ευρώπη και υπάρχουν και ενδιασμοί εκ μέρου πολλών για τον τρόπο με τον οποίο ενεργούν οι κυβερνήσεις τους, σε ποιο συμπέρασμα καταλήγω. Ότι πολλοί θέλουν περισσότερη Ευρώπη την ώρα της αλήθειας. Δεν θέλουν, αλλά σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα πιστεύω ότι όλοι οι συντάκτες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι χρειαζόμαστε περισσότερο Ευρώπη. Γι' αυτό προτείνουμε εμείς για τέτοιου είδου θέματα, αμυγό ευρωπαϊκά, να έχουμε περισσότερη βρώμη. Συγγνώμη, πριν να τελειώσω κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα για τεχνικούς λόγους να πω το εξή. Οι τροπολογίες συμπεριλαμβάνονται σε τέσσερα διαφορετικές εκθέσεις, δεδομένου ότι αφορούν τέσσερις διαφορετικές εκθέσεις ε, της ΕΚΟΝ. Εγώ προσπάθησα με διάφορες αποχρώσεις διαφορές το θέμα αυτό να το εξετάσω διεξοδικά και επαναλαμβάνω τις έχετε εδώ όλες τις τροπολογίες τις δικές μου και βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας για την ε, μοίρα τους. ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα σαν Θεμέντες Νεβίγκο. Πάρα πολύ σοβαρή, εντατική δουλειά που κάνετε συνθετική και με τα διαγράμματα και με τα slides και με την γλαφυρή παρουσίαση που μας προσφέρατε. Ο κύριος Βέροστατ πρώτος έχει το λόγο. Βέροστατ. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Μέντες Ντεβίγκο για <clears throat> την παρουσίασή του, για την τις εξηγήσει του, την έκθεσή του και σαν νομικός και σαν συνταγματολόγος θα ήθελα να ξέρω πώς ε, ασχολήθηκε τώρα με τα οικονομικά. Είναι μια ε, νέα στροφή στην καριέρα του. Το βασικό όμως είναι ότι περισσότερες τροπολογίες τις οποίες ε, έχει εκπονήσει με τους τέσσερις εισηγητές της Επιτροπής Οικονομικών είχαν, είχαν εξετάσει την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά προχώρησαν πέραν των προτάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ουσιαστικά και ίσως θα προσπαθήσω να συνοψίσω ασχοληθήκανε με τον ρόλο και την ισχύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πράγμα το οποίο προκύπτει, το οποίο οδηγεί σε διάφορες τροπολογίες και μετά εξετάζει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής όσον αφορά τη διάστασή της, τη δομή της και τρίτον και μετά στο αρμπιτράζ το οποίο αναφέρεται εδώ διότι Δε, όταν υπάρχει μία διαφορά μεταξύ των διαφόρων εθνικών αρχών διότι ε, όπως είπα και στους τέσσερις εισηγητές της Επιτροπής ΕΚΟΝ ε, συγχαίρω, συμφωνώ και ε, εφόσον έχουν συνεννοηθεί με τον κύριο ο Μέντες δεν θα προχωρήσουμε ε, πέραν των προτάσεων του Συμβουλίου επανερχόμαστε στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αν συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο τόσο καλύτερο διότι όσο πιο ισχυρό εμφανίζεται το Κοινοβούλιο τόσο περισσότερα επιχειρήματα θα έχουμε στην διαιτησία με το ε, Συμβούλιο, διότι ε, θα πρέπει να ε, εκπονήσουμε τροπολογίες, θα υπάρξει μάχη και εμείς πρέπει ε, να ε, θεωρήσουμε σημείο κινήσεώς μας ε, την ευρωπαϊκή πρόπτικη που πρέπει να καλύψει η πρόταση της Κομισιόν. Λοιπόν, κύριε Μέντες Βουίγκο, μόνο ένα ασθενές σημείο υπάρχει, το οποίο είναι το εξής. δεν φτάσαμε στην ε, τελική ε, κατάληξη, δηλαδή να υπάρξει μόνο μία αρχή, θα έχουμε τέσσερις αρχές. Μία για το συστηματικό κίνδυνο, δηλαδή μακροπρόθεσμη εποπτεία, η έκθεση της κυρίας Γκουλάρ και μετά οι τρεις μικροαρχές. αρχές. Την προηγούμενη φορά το είχα ήδη πει στον κύριο Μέντες Ντεβίγκο. Ουσιαστικά θα έπρεπε να απλοποιήσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά πρέπει να ξέρουμε κύριε Πρόεδρε ότι οι συγητές της Επιτροπής Οικονομικών θεώρησαν ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον διότι είχαν προτείνει οι τέσσερις αρχές, η μία μακροοικονομική αρχή και οι τρεις μικροοικονομικές ε, να συνεργάζονται, να υπάρξει ένα joint committee, μία κοινή επιτροπή και να καταλήγαμε σε πέντε. Μία μακροοικονομική, τρεις μικροοικονομικές και μία κοινή επιτροπή η οποία θα συντόνιζε ε, τις τρεις μικροοικονομικές ε, αρχές. Θα χρειαζόμαστε το συντονισμό. Τέλος πάντων. Καταλήγοντας όμως, όλοι οι συγητές είπαν ότι όλα τα όργανα αυτά έπρεπε να είναι σε ένα σημείο. Θα πρέπει λοιπόν να προτείνουμε να υπάρξουν τέσσερις ε, οργανώσεις και μία κοινή επιτροπή που θα συνεργάζονται στενά. Νομίζω ότι είναι ένας πρακτικός τρόπος ε, με τον οποίο λέμε ότι τουλάχιστον ε, στην ενδιάμεση αναθεώρηση, την mid-term review η οποία προτείνεται, όλα αυτά μπορούν να συγχωνευτούν σε ένα σύστημα και θα έχουμε μία αρχή για τις τράπεζες, μία ε, για το ασφαλιστικό σύστημα, μία για την περίθαλψη αλλά και μία για τα χρηματοοικονομικά παράγωγα. Ε, δηλαδή θα υπάρχει ε, ε, ένας που θα συντονίζει όλους τους άλλους και θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να ξεχωρίζουμε την μακροπρόθεσμη προοπτική από την μάλλον τη μακροοικονομική προοπτική από την μικροοικονομική και θεωρώ ότι καλό είναι να γνωρίζουμε και σε μικροοικονομικό επίπεδο τους κινδύνους που προκύπτουν μακροοικονομικά Υποθέτω όμως ότι οι αρχές δεν κατάφεραν να υιοθετήσουν αυτή τη λογική, δηλαδή όλα να περιληφθούν σε μία αρχή τις συντάξεις, ε, τις ασφάλειες, ε, τις τράπεζες και τότε οι, ε, οι συγητές μας είπαν τουλάχιστον τέσσερα όργανα αλλά στο ίδιο σημείο με έδρα στη Φραγκφούρτη που θα ήταν μια εγγύηση ότι ίσως σε δυόμιση χρόνια θα μπορέσει να υπάρξει συγχώνευση μιλάμε για mid-term review, για ενδιάμεσο απολογισμό. Όσον αφορά τώρα α, τους εισηγητές θεωρούσαν ότι είναι καλύτερα να υπάρξουν ε, τέσσερις οργανώσεις σε ένα σημείο αντί ε, για τρία σημεία, δηλαδή αν μία ήταν στο Λονδίνο, η άλλη στο Παρίσι, η άλλη στη Φραγκφούρτη και κύριος είδεν πού η τέταρτη, για να είναι όλα τα κράτη ευχαριστημένα θα είχαμε τρεις έδρες και ε, η μία αρχή ε, για τη συντάξη θα ήταν σε ένα μέρος και διαφορετικά μια άλλη υποδιέρεση θα μπορούσε να είναι κάπου αλλού αλλά νομίζω τελικά καλά έκαναν οι νομοθέτες και είπαν θα επικεντρωθούμε σε ένα ε, γεωγραφικό σημείο κατά τρόπο ώστε στα επόμενα έτη να μπορέσουν να συγχωνεύσουμε όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Δεν ξέρω μέχρι πότε υπάρχει προθεσμία για τροπολογίες, αλλά ίσως με τον κύριο Μέντες Δεβίγκο και τουλάχιστον με τη βοήθεια των τριών από τους τέσσερις εισηγητές Πιστεύω όμως ότι τρεις από τους τέσσερις εισηγητές θα συμφωνούσαν να μπορέσουμε να ξανασκεφτούμε το όλο θέμα και να δούμε μήπως μπορούμε να προχωρήσουμε ε, πιο ριζικά. Δηλαδή, ε, όταν ε, υπάρξουν σαν διαπραγματευτική θέση οι τέσσερις αυτές ενότητες εις ένα γεωγραφικό σημείο ως έδρα, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, μία αρχή δηλαδή, ένα ε, διευθυντήριο ή κατά τη γνώμη μου και ε, μία αρχή με ε, μία διεύθυνση μακροοικονομίας και άλλες τρεις μικροοικονομίες. Τέλος πάντων έχουμε ακόμη χρόνο, δεν πρέπει να βιαστούμε, και θα πρέπει και ο κύριος Μέντες Δεβίγο και οι άλλοι εισηγητές να μπορέσουν ίσως να καταλήξουν σε μία τροπολογία για μία αρχή με τρία-τέσσερα διευθυντήρια αντί για τέσσερις οργανώσεις οι οποίες θα εδρεύουν σε ένα κοινό σημείο π.χ. τη Φραγκφούρτη. Ε, το συζήτησα με την κυρία Γκολάρ και με τους άλλους συζητητές και νομίζω ότι έτσι θα έχουμε μια πολύ πιο ισχυρή διαπραγματευτική θέση από ότι αν συμφωνήσουμε εκ προημίου και πούμε ότι εντάξει θα υπάρξει αυτή η ε, δομή των τεσσάρων ε, χωριστών αρχών. Ε, πιστεύω ότι ο κύριος Μέγκας Βίγκο έχει κάνει ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση με την έκθεσή του και ε, όταν θα έχουμε το τελεσίδικο κείμενο ε, θα καταρτήσουμε τροπολογίες και ενδεχομένω θα προχωρήσουμε και περισσότερο. Ίσως δεν είναι ακριβώς αυτό που ήθελε το Συμβούλιο, αλλά ίσως μπορέσουμε να προχωρήσουμε και πέραν από αυτό το οποίο ε, επιθυμούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν υπέβαλε την πρόταση το Σεπτέμβριο. Στις επόμενες εβδομάδες ή στον υπολοιπόμενο χρόνο μέχρι ισότου κατατεθούν οι τροπολογίες πρέπει να δούμε αν θέλουμε να προχωρήσουμε περισσότερο. Κατά τα άλλα, υπάρχουν ορισμένες ε, λεπτομέρειες ε, ε, στις τροπολογίες που πρέπει να εξεταστούν αν θα μιλάμε για οθόρητη ή οθόρητης ε, πληθυντικό ή όχι και τέλος ε, ε, και πάλι συγχαίρω τον κύριο Μέντες Δεβίγκο για την εργασία του καταλήγει να είναι ένας οικονομολόγος και ειδικό. Ας δώσουμε δώσα ε, λίγα λεπτά. Ε, θέλω να ευχαριστήσω τους διερμηνείς που μας διέθεσαν πέντε λεπτά ακόμη για να δώσουμε τη δυνατότητα στον κύριο Μέντες Δεβίγκο να απαντήσει ε, και θα πρέπει να καθορίσουμε και την προθεσμία για τις τροπολογίες 7 Απριλίου για να έχουμε καιρό να το σκεφτούμε. 11 Μαρτίου. Μεντές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Βερχοφστάτ για την παρέμβασή σας. Όντως, οι προτάσεις των τεσσάρων συναδέλφων και οι τροπολογίες είναι παρεμφερείς με αυτά που θα συζητηθούν αύριο στην ΕΚΟΝ. Γιατί, Γιατί εγώ το θέμα αυτό το συζήτησα από κοινού με τους συναδέλφους της Επιτροπής ΕΚΟΝ και πρέπει να σας πω ότι τα αποτελέσματα όλη αυτή τη δουλειά για μένα είναι πάρα πολύ ικανοποιητικά. Εγώ το θέμα που ανέφερε ο κύριος Βέρχοφ Στάτη ήδη το είπα την ε, ε, τελευταία φορά ότι ίσως για τις τρεις ε, μικροοικονομικές αρχές να κάνουμε μία. Αλλά μου φαίνεται ότι οι κύριοι εισηγητές δεν ήταν ε, σύμφωνη, γι' αυτό την εγκατέλειψα. Πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι αύριο θα έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε τα θέματα αυτά στην ε, Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων αύριο το απόγευμα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη συζήτηση και μετά θα μπορέσουμε να συναντηθούμε ε, οι εισηγητές και εγώ και όποιον ενδιαφέρεται από την Επιτροπή να έρθει να το συζητήσουμε τα όλο θέμα, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα θέμα που χρειάζεται να μελετήσουμε διεξοδικά. Πιστεύω ότι θα πρέπει να καθορίσουμε με μια κατάθεση τροπολογιών διότι ίσω θα μπορούσαμε να δώσουμε κάποιε ιδέε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Το έχουμε κάνει αυτό και νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε. Διότι ό,τι και να κάνουμε θα είναι μια κάποια προστιθέμενη αξία. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι εσείς προτείνετε έχει καλός για μένα. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 15 Μαρτίου. Έχει καλός. Έχουμε σχεδόν ένα μήνα στη θέση μας. Νομίζω ότι είπατε 15 Μαρτίου, δεν είναι έτσι. Και μετά θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Βέρχοφστατ, το οποίο βλέπω ότι, είναι, ότι την ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα, ή όποιον άλλο θέλει να έρθει σε επαφή μαζί μου για να το συζητήσουμε ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε πραγματικότητα αυτό που όλοι πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να γίνει την ε, παύριο της οικονομικής κρίσης και Έχω την εντύπωση ότι όπως σας είπα αυτό που κάνουμε σήμερα είναι ως λύση μια αποκορυφωμένη λύση. Δεκαφεϊνέ όπως είπα στην αρχή. Θα πρέπει όμως τη στιγμή που υποβάλλουμε προτάσεις να υποβάλλουμε προτάσεις δημιουργικές για να αποδείξουμε ότι και με τη συνθήκη της Λισαβόνας κερδίσαμε σε αρμοδιότητες και χρησιμοποιούμε αυτή το προνόμιο. Και βεβαίως ότι προτισκάνουμε να την κάνουμε με συνεχτικό τρόπο. Θα ήθελα να πω στη, λοιπόν ότι εγώ θέλω να πούμε κάτι το οποίο θα είναι συμπληρωματικό σε αυτά που λέει η ΕΚΟΝ και να βοηθήσει τις αποφάσεις της ΕΚΟΝ βεβαίως στα πλαίσια πάντων ορμοδιοτήτων μας και πάντα στα πλαίσια της συνθήκης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Βερχοφστάτ, ευχαριστώ τον κύριο Βντεβίγκο. Είχα μιλήσει για τις 11 Μαρτίου, δεν κάνω λάθος, και το ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 7 Απριλίου. Αυτά, δεν έχω καμία άλλη ανακοίνωση να κάνω. Λύεται η συνεδρίαση. Ευχαριστώ και εσάς και τους διερμηνείς. Υπενθυμίζω ότι η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 17 και στις 18.